Okay, good morning, friends. Λοιπόν, καλημέρα σας αγαπητοί φίλοι. Morgen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, άρχεται η συνεδρίαση μας πάλι που είχε διακοπεί χθες το απόγευμα δεν ξέρω τι συνηθίζεται εδώ, αλλά λόγω της βεβαρημένης ημερησίας διάταξης θα ήταν καλό να αρχίσουμε στην ώρα μας. Περνάμε στο σημείο 8 της ημερησίας διάταξης, απαλλαγή για τα άλλα θεσμικά ε, όργανα. Η συγγήτρια είναι στα σέντρα. Ο Λούι Γκαλέα από το Ελεκτικό Συνέδριο είναι εδώ και θα ήθελα να τον παρακαλώσω να μας κάνει την παρουσίασή του. Παρακαλώ κύριε Γκαλέα, έχετε το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλα τα αξιότιμα μέλη και τον διακεκριμένο Δόκτωρα Σόλτς που είναι εδώ παρόν όπως θα το έχετε συνηθίσει κι εσείς όταν συζητά την απαλλαγή αυτή η Επιτροπή των άλλων οργανισμών, των άλλων θεσμικών οργάνων πρέπει να γίνεται αναφορά στο κεφάλαιο 7 της ετησίας εκθέσεως του ελεκτικού συνεδρίου όπου εκεί παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα ειδικών αξιολογήσεων διοικητικών δαπανών των θεσμικών οργάνων και άλλων οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ενώσης. I think it uh, uh, Είναι σημαντικό πιστεύω να ξεκαθαρίσουμε κάτι ότι το ελεκτικό συνέδριο κάνει μια γενική αξιολόγηση όσον αφορά τις δικαιτικές δαπάνες για όλα τα θεσμικά όργανα και άλλους φορείς ε, ομού. Επί της βάσεως δοκιμών τυχαίου δείγματος συνολικού συναλλαγών που καλύπτει όλο τον τομέα αυτών. Ε, τα αποτελέσματα των ελόγων αξιολογήσεων για το οικονομικό έτος 2010 ε, είναι θετικό και το ελεκτικό συνέδριο μπόρεσε να συμπεράνει ότι οι συναλλαγές που δημιουργούν στις δαπάνες το 2010 από κάθε ηλική άποψη ήταν συναλλαγές τακτικές και νόμιμες. Αυτό συμφωνεί και με πρώτερα έτη. Το ελεκτικό συνέδριο, όπως προανέφερα, παρέχει γνωμοδότηση για όλα τα θεσμικά όργανα και άλλους φορείς. Εν γέννη, και δεν δίνει ξεχωριστή γνωμοδότηση για κάθε ξεχωριστό θεσμικό όργανο ή φορέα. Όμως το ελεκτικό συνέδριο κάνει και άλλες εργασίες, ούτως ώστε να μπορέσει να παρουσιάσει ε, κάποιες παρατηρήσεις επί κάποιων φορέων. Αυτή η συμπροματική δουλειά έχει σαν στόχο συγκεκριμένα θέματα, επιλεγμένα θέματα. Σε αυτή την περίπτωση επιλέξαμε να κάνουν περαιτέρω εργασίες επί υπολογισμού και πληρωμής αποζημιώσεων συντάξεων μισθών ε, και διαφόρων δαπανών που αφορούν διαδικασίες προσλήψεων, ε, μονίμου προσωπικού, προσωπικού επισυμβάση, προσωρινού προσωπικού και επί διαφόρων συμβάσεων προμηθειών. Η φετινή έκθεση για το 2010 συμπεριλαμβάνει και σχόλια. Αυτά αφορούν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, οι παρατήρησει του ε, ελεκτικού συνεδρίου αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ε, καλύφθηκε η οικοδόμηση του κτηρίου Residence με μεταφορές από κονδύλια από άλλους τομείς αντίθετα με την αρχή της ε, δημοσιονομικής ακριβίας. Όσον αφορά την ΟΚΕ, το ελεκτικό συνέδριο σχολίασε ότι η σαν μέθοδος για την αποζημίωση οδηπορικών, για τα μέλη αυτής, δεν ευθυγραμμίζεται με τη βάση ότι τα οδηπορικά θα πρέπει να αποζημιώνονται επί τη βάση των πραγματικών ε, δαπανών. Το ελεκτικό συνέδριο επίσης ε, σημείωσε δυναμίες όσον αφορά τις διαδικασίες προμηθειών. Τώρα όσον αφορά την Επιτροπή των Περιφερειών, το ελεκτικό συνέδριο ενετόπισε αδυναμίες όσον αφορά τη διαδικασία προμηθειών, όσον αφορά τις διαπραγματευτικές ε, διεργασίες. Και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων, σημειώνει το Ελεκτικό Συνέδριο ότι αυτή η υπηρεσία κάλυψε κάποια κενά από τη βάση εσωτερικών διαγωνισμών όταν οι βέλτιστες πρακτικές θα έπρεπε να επιβάλλουν την χρήση των υπηρεσιών της ΕΠΣΟ. Στην ετήσια έκθεσή μας επίσης σχολιάζουμε τις εξελίξεις που αφορούν τις συστάσεις που έγιναν σε πρώτερες εκθέσεις μας. Ένα από αυτά αφορά την Ευρωπαϊκή υπηρεσία, Εποπτική, Υπηρεσία Προστασία των Δεδομένων, όσον αφορά την καταβολή ε, των διαφόρων κοινωνικών επιδομάτων στα μέλη του προσωπικού. Συστήσαμε ότι σε κάποια χρονικά διαστήματα θα πρέπει το προσωπικό να παρουσιάζει έγγραφα, θα επιβεβαιώνουν ποια είναι, η κατάστασή του η προσωπική. Σημείωσε το ανοιχτικό συνέδριο μέσα που εισήχθησαν για να καλυφθεί, θεσπίστησαν μάλλον, να καλυφθεί αυτό το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την προσοχή σα, ευχαριστώ και τα μέλη τη επίτροπή και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκαλία. Πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, θα ήθελα να καλωσορίσω τώρα τους εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων από το Ελεκτικό Συνέδριο, τον κύριο Βίθ Καρσία, από το δικαστήριο. Αλφρέδο, Αλφρέδο, Αλφρέδο Καλότ. και τον κύριο Στάλ από την Επιτροπή των Περιφερειών, τον κύριο Βεστλάκε από, το, ε, από την ΟΚΕ, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τον κύριο Ντόξη από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εποπτείας της Προστασίας των ε, Δεδομένων και από τον Βάτα τον κύριο Χάρντεν. Καλώς ορίσατε όλοι και θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην εισηγήτρια του τόσο σημαντικού αυτού θέματος. Η κυρία Γιάλα Σέντερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας συγχαρώ θερμότατα για τον ορισμό σας ε, στη θέση του Πρόεδρου της Επιτροπής μας. Ελπίζω να έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία. Η Επιτροπή μας άλλωστε ασχολείται με θέματα συναισθηματικά φορτισμένα λιγότερο ή περισσότερο, αλλά αυτό που σίγουρα πρέπει να κάνουμε είναι να εργαστούμε για να βελτιώσουμε τα τη λογιστική διαχείριση και απέναντι στην κοινή γνώμη και στους πολίτες. Ακούσαμε λοιπόν την ομιλία του εκπροσώπου του ελεγκτικού. Θα έχουμε και μία πρώτη ε, δραστηριότητα αυτή τη στιγμή, δηλαδή η ακρόαση των υπευθύνων διαχείριση σε διάφορα θεσμικά όργανα πλήν του Συμβουλίου στο πλαίσιο του ελέγχου των λογαριασμών των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Και ευχαριστώ τους παρισταμένου εδώ που θα μας δώσουν τις πληροφορίε που μας είναι απαραίτητες για να ολοκληρώσουμε τις δικές μας εργασίες. Πρώτα απ' όλα όμως θέλω να σας παρακαλέσω κύριε Πρόεδρε να δώσουμε σε καθέναν από τους ε, παρισταμένου τη δυνατότητα να μας κάνουν μια σύντομη παρουσίαση ολιγόλεπτη να ακούσουν όλοι οι παρόντες ε, τα σχετικά με το κάθε θεσμικό όργανο και μετά θα κάνω εγώ τις ερωτήσεις μου και βέβαια και οι συναδελφοί μου μπορούν ε, να, ε, θέσουν τα ερωτήματά τους. Ήδη έχουν υποβάλει εγγράφους ερωτήματα και τους ευχαριστώ για τη συνεργασία τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή που μα κάνατε. Και ναι, θα ακολουθήσουμε αυτή την πρόταση που κάνατε. Καταρχήν θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Καλώτη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Παρακαλώ. Monsieur Καλώτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι αρκετά σύντομος και λακωνικός. Ικανοποιηθήκαμε προφανώς από την αναφορά που έγινε από πλευράς ελεκτικού συνεδρίου στην ε, έκθεση. Δεν έκανε καμία παρατήρηση όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, άρα είμαστε ικανοποιημένοι. Διότι κατά κάποιο τρόπο βλέπουμε τους καρπούς εργασιών προσπαθίας που καταβάλαμε επί σειρά ετών όσον αφορά την συνεργασία με το ελεκτικό συνέδριο όσον αφορά τον ετήσιο έλεγχο και συνεργαστήκαμε και με άλλε ελεκτικέ αρχέ και όλου ιδιαίτερω με την Επιτροπή Δημοσιονομικού ε, Ελέγχου του Προλογισμού, μάλλον. Αυτό το κάναμε για να προσπαθήσουμε να δώσουμε τι πληρέστερε πληροφορίε όσον αφορά τι δραστηριότητέ μα. Έτσι το καταφέραμε. Ε, και από την άλλη προσπαθήσαμε να λάβουμε πλήρω υπόψη τα σχόλια και τις προτάσεις που εμπεριέχονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει της εκθέσεως της ε, Κοκομπή. Όσον αφορά τους ελέγχους, περιορίζουμε σε αυτό που λέω, όσον αφορά τις θηριότητες του θεσμικού οργάνου, θα δείτε τις δραστηριότητε του 2010, ότι εκεί θέλαμε να υπογραμμίσουμε την εντατικότητα των διαφόρων ε, ε, δραστηριοτήτων του ελεκτικού συνεδρίου των τριών φορέων αυτού με δείχνουν αύξηση των υποθέσεων κάθε χρόνο και μπορώ να σας πω ότι αυτή η αύξηση των υποθέσεων αντικατοπτρίζεται και στα στοιχεία του 2011 που εξετάζουμε και που θα δείτε σύντομα και πριν από ότι το 2011 μπορέσαμε να χειριστούμε αυτή τη ροή των υποθέσεων αλλά η ανησυχητική κατάσταση, ιδιαίτερα όσον αφορά το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενώσεω από τα τρία δικαστήρια που παρτίζουν το όργανο, οδήγησε το Μάρτιο 2011 να υποβάλει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο μια πρόταση τροποποίησεως ε, του καταστατικού του ε, για να ενισχυθεί η δυνατότητα που θα έχει το δικαστήριο για να αντιμετωπίσει το φόρτο εργασίας με αλλαγές που αφορούν τη σύνθεση του δικαστηρίου και των αντιπροέδρων για να υπάρξει καλύτερη διαχείριση των εκδικάσεων και όσον αφορά το δικαστήριο να προσθεθούν 12 νέοι δικαστές για να αντιμετωπιστεί αυτή η αύξηση ανησυχητική του ρυθμού των υποθέσεων. Υπάρχει ένα στοιχείο που αφορά τις δραστηριότητε που ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σωστά. Είναι η διάρκεια των υποθέσεων, εκδικάσεων των υποθέσεων και όσον αφορά το δικαστήριο και τις προδικαστικές υποθέσεις, παραπομπές, που είναι κάτι πολύ σημαντικό όσον αφορά τις εργασίες μας και ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η διάρκεια των υποθέσεων ήταν 24 μήνες το 2004 και πήγε 16 μήνες το 2010 και παραμένει στους 16 μήνες το 2011 παρά την αύξηση των αριθμών των προδικαστικών ε, υποθέσεων. Άρα μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι, πιστεύω, στο δικαστήριο, αλλά έχουμε και λόγου για να λάβουμε νέα μέτρα και άλλα μέτρα που θα επιτρέψουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να συνεχίσει να εκπληρώνει την αποστολή του σωστά στο μέλλον, ε, στο πλαίσιο που σας ε, περιέγραψα. Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Ε, Ευχαριστώ κύριε Καλότσο. Νομίζω θα ήταν λογικό να ακούσουμε όλα τα θεσμικά όργανα και μετά να έχουμε τις απαντήσεις. Επόμενος εξονόματος του Συνελεκτικού Συνεδρίου, ο κ. Ζουίθ Καρσία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψατε μου και εγώ να σας συγχαρώ πρώτα απ' όλα για τον πρόσφατο ορισμό σας. Εν συντομία θα ήθελα να επισημάνω τα σημαντικότερα στοιχεία της διαχείρισης του ελεγκτικού συνεδρίου κατά το οικονομικό έτος 2010. Πρώτα απ' όλα να πω ότι το 2010 επιβεβαιώθηκε η βελτιωμένη αποτελεσματικότητα του συνεδρίου. 62 έγγραφα ε, συν 4 σε σχέση με την προηγούμενη δουλειά. Δηλαδή, εκπονήσαμε μεταξύ των οποίων 14 ειδικέ εκθέσει. Πρόκειται για μια τάση η οποία μεταφράστηκε και σε μια θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά του βασικού δείκτε ε, αποτελεσμάτων και performance indicators και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση τη ποιότητα των εκθέσεών μα ε, και την αποδοχή των συστάσεών μα. Οι δείκτε δείχνουν βέβαια παρόλα αυτά ότι πρέπει να βελτιωθούμε σε δύο σημαντικού τομεί αυτό το αναφέρει και η ετήσια έκθεσή μας. Συγκεκριμένα η ακρίβεια και στις εκθέσεις ε, αλλά και στην ε, κοινοποίηση των ε, πορισμάτων μας προς τους ελεγχθέντες. Το συνέδριο προσπάθησε να προβεί σε μια αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του. Το ποσοστό τη δημοσιονομική εκτέλεση, εκτέλεση του υπερπολογισμού σε σχέση με το προηγούμενο Έτο βελτιώθηκε, 93% είναι το ποσοστό αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά τι κενέ θέσει μειώθηκαν σημαντικά. Το 2010 ήταν κάτω από το 5% αυτό το ποσοστό και μπορώ να σα πω ότι αυτή τη στιγμή ε, είναι γύρω στο 3%. Επίσης, 26 ε, θέσεις διοικητικές ε, μεταφέρθηκαν στο Core business, ε, στις ε, θέσεις των ελεκτών δηλαδή, μια τάση που δεν θα περιοριστεί μόνο στο 2011 αλλά και στα επόμενα χρόνια ε, θα το έχουμε το ίδιο το στοιχείο αυτό. Επίσης κάναμε σημαντικές εξοικονομίες το 2011. 500.000 ευρώ ετησίως στις υπηρεσίες ασφάλειας και υποδοχής και πάνω από 120.000 ευρώ ετησίως υπηρεσίες καθαριότητας. Τέλος, το σχέδιο για το κατ' 3 το νέο μας κτίριο, προχωρά σύμφωνα με το προεπόμενο χρονοδιάγραμμα, χωρίς να έχουμε υπέρβαση του κόστους που περιλάβαμε στον προπολογισμό. Θα ήθελα να πω ότι το 2010 ε, δείξαμε ως συνεδριό ότι μας ενδιαφέρει να ε, δείχνουμε ευθύνη, υπευθυνότητα και το ε, έδειξε αυτό και η θετική υποδοχή των εκθέσεων και τα σχόλια του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ήταν θετικά σε σχέση με τα διάφορα σχέδια προπολογισμού τα οποία επέβλησαν τα τελευταία χρόνια. Τέλος, είχαμε και θετικές εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελεγκτή. Εν κατακλείδη, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι το 2010 ήταν μια χρονιά που οι προσπάθειες εξυγχρονισμού του συνεδρίου συνέχισαν να δίνουν καρπούς, προσπάθειες που θα συνεχιστούν η δημοσιονομική κρίση μας υποχρεώνει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, δηλαδή να παράγουμε περισσότερες ε, εκθέσεις αλλά και με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και επίσης να κάνουμε και μεγαλύτερη ε, οικονομία, να περιορίσουμε τους ήδη περιορισμένους ε, πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Άρα πρέπει να βελτιώσουμε καλύτερα την οργάνωση των εργασιών μας και την παραγωγικότητά μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν, δρομολογήσαμε αρκετές πρωτοβουλίες, μία εξ αυτών είναι η, το peer review εξελέγηση από ομοτήμους. Θα ξεκινήσει φέτος και θα συνεχιστεί αυτό το εγχείρημα και θα ενημερώνουμε το Κοινοβούλιο. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ουρίθ Καρθία. Ο Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής των Περιφερειών έχει τώρα το λόγο. Ο κύριος Σάλ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Επιτροπή των Περιφερειών το περασμένο έτος προσπάθησε να βελτιώσει τις ε, διοικητικές της δραστηριότητες. Βέβαια, ε, ακολουθώντας τις ενδείξεις του ηλεκτρικού συνεδρίου και τι ενδείξει που πήραμε στο παρελθόν κατά τη διάρκεια των διαδικασιών απαλλαγή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά τα στοιχεία ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Εισαγάγαμε μια διαδικασία αυτοελέγχου όπως την είχε αναπτύξει στο παρελθόν το Διοικητικό Συνέδριο και έτσι μπορέσαμε να εξυγχρονίσουμε το διοίκησή μας, πράγμα που συνεχίζουμε να κάνουμε και που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί με τη συνθήκη της Λισαβόνα η Επιτροπή των Περιφερειών αποκτά σε περισσότερες αρμοδιότητες και καλούμεθα να χρησιμοποιούμε τους πόρους μας κατά δυνατόν ε, οικονομικά και αποτελεσματικά. Δεν θέλω να σας ε, απαριθμίσω τώρα που θα πρέπει ακόμα να βελτιώσει τη διαστηριότητά της η Επιτροπή των Περιφερειών αλλά να σας πω και όσον αφορά τις νομοδοτήσεις και όσον αφορά την έκθεση δραστηριότητα μας θα πρέπει να είμαστε πιο ε, αποτελεσματικοί και ήθελα να πω ότι μέσα στα πλαίσια της Ένωσης για την ε, Μεσόγειο ε, παρεκλήθη η Επιτροπή των Περιφερειών από τις κυβερνήσεις να συντονίσει τη συνεργασία των τοπικών διοικήσεων της ε, περιοχής της ε, Μεσογείου. Αυτό συνενώντας και ε, προσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τοπικούς εκπροσώπους. Πρέπει και εκεί δηλαδή να δράσουμε. Για να αναφερθώ τώρα στα θέματα που τίθενται μέσα στα πλαίσια της έκθεσης του ηλεκτρικού συνεδρίου, θα ήθελα να σας πω ότι μέσα στα πλαίσια των διαγωνισμών με χαμηλό ποσό υιοθετήσαμε διάφορα μέτρα ούτως ώστε να βελτιώσουμε την ε, ε, συνεργασία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών. Κάτω τα άλλα, ετέθησαν και άμεσες ερωτήσεις προς τα θεσμικά όργανα. Θα μπορούσα ίσως σύντομα να αναφερθώ στις ερωτήσεις αυτές. Θέλετε να αναφερθώ στις ερωτήσεις αυτές κύριε Πρόεδρε τώρα. Πρόεδρος, κοιτάξτε, στα σύντομα να αναφέρετε τα σημεία που θεωρείτε πάρα πολύ σημαντικά εσείς ο ίδιος. Äh, äh, άρα νομίζω ότι παρουσίασα στα σύντομα την θέση Επιτροπής των Περιφερειών και κατέδειξα ότι εμείς προσπαθούμε με λίγους πόρους να τοποθετούμε έτσι ούτως ώστε να δρούμε αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Πρώτος ευχαριστώ κύριε Στάλ. Επόμενος, ο Γενικός Γραμματέας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ο κύριος Βέστιλακ, παρακαλώ. Thank you very much. Um, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, για τις, κρατικές, για τις ε, δημόσιες προμήθειες, η Επιτροπή σημείωσε δεόντως τις παρατηρήσεις του ελεκτικού συνεδρίου. Επεστάλλει υπενθύμηση σε όλου του υπεύθυνου για διοδότηση ε, με ανάθεση στο πλαίσιο αυτό και προσπάθησε να επισημοποιήσει η Επιτροπή περαιτέρω την ομαδοποίηση τέτοιων πόρων, ούτω ώστε να σεβαστούμε πλήρω τι παρατηρήσει του ελεκτικού συνεδρίου. Όμω, Αναγνωρίζω ότι μικρότερα θεσμικά όργανα έχουν κάποια δυναμία σε αυτό το τομέα, διότι έχουν περιορισμένη ομάδα ανθρωπίνων πόρων ε, εν πρώτης. Και γι' αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερως η επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου που έλαβα, όπου είπε ότι ίσως ε, τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο για να συνεργαστούν σε διάφορους τομείς και στις δημόσιες προμήθειες και αυτό είναι κάτι στο οποίο προσβλέπω να το συζητήσω με τους διάφορους συναδέλφους γενικούς γραμματείς όσον αφορά την απαλλαγή του 2009 και τη σχετική διαδικασία και τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο πρόεδρος Νίλσον έγραψε στον πρόεδρο Μπούτσεκ στις 24 του Οκτωβρίου πέρσι με λεπτομερή απάντηση σε όλες τις συστάσεις που έκανε το Κοινοβούλιο σε αυτό το πλαίσιο και δεν θα επαναλάβω τα περιεχόμενα της επιστολής, είμαι σίγουρος ότι ε, τα έγγραφα τα έχετε Πανερχόμενο στι παρατηρήσει του ελεκτικού συνεδρίου υπήρξε και κάποια παρατήρηση που ανέφερε ο Δ. Γαλέα στην παρουσίασή του όσον αφορά ε, το οικονομικό καθεστώς των μελών της Επιτροπής. Εκεί με τα χαράς ενημερώνω τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ότι στις 6 Δεκεμβρίου πέρσι το Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Οικονομική και Κοινωνικής Επιτροπή ομοφόνο απεφάσισε να απαλλαγεί με την επιλογή κατά αποκοπή που προβλέπεται και να αντικαταθεί με ένα σύστημα που συνάδει με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα σύστημα που βασίζεται κατά πολύ στο σύστημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βασικά στοιχεία των λόγων συστήματος συμπεριλαμβάνουν τις αποζημιώσεις που θα καταβάλλονται επί πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στα αυτά τα ταξίδια και οροφή για τα εισιτήρια business και να ευθυγραμμιστούν οι μερικές αποζημιώσει με τις τη Επιτροπή των Περιφερειών και τα διπορικά να είναι παρόμοια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Εδώ θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να χαιρετήσω τις συμβουλές που λάβαμε από τον ε, εισηγητή για την απαλλαγή του 2010 σχετικά με το θέμα. Όσον αφορά τις ε, καθημερινές αποζημιώσεις, είναι ανομαλία ιστορική το ότι ο ΚΕ αντίθετα από την Επιτροπή των Περιφερειών χρειάζεται τη συμφωνία του Συμβουλίου των Υπουργών ούτως ώστε να αλλάξει τις ε, καθημερινές αποζημίες των μελών. Σήμερα είναι 233 ευρώ την ημέρα, συν 34 ευρώ, 34 επαναλαμβάνω ευρώ, αν τα μέλη πρέπει να διανυχτερεύσουν. λαμβάνοντα υπόψη ότι τα μέλη τη Επίτροπή των Περιφερειών δεν έχουν ευρωπαϊκού μισθού. νομίζω ότι τα αξιότιμα μέλη θα συμφωνούν ότι είναι και ώρα οι αποζημιώσει να ευθυγραμμιστούν περισσότερε αποζημιώσει Επιτροπή των Περιφερειών που αυτόνομα καθορίζει τι καθημερινέ αποζημιώσει και έχει εξασφαλίσει το ότι παραμένουν, επιτρέψτε μου να πω, οι αποζημιώσει ρεαλιστικέ. Σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θα ελπίζαμε ε, να μας δει με δίκαιο όμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της απαλλαγής ώστε να πιστεί το Συμβούλιο να αλλάξει τις καθημερινές, ε, ε, την εμείς αποζημίωση των μελών. Συνοψίζοντας όσον αφορά τις δύο παρατηρήσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου η Επιτροπή έκανε σημαντικά βήματα και όσον αφορά την απαλλαγή του 2009 και τις σχετικές συστάσεις, η Επιτροπή εξίσου έλαβε δεόντως υπόψη τα σχόλια και έκανε σημαντικά βήματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενο ομιλητή για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, ο κύριο Σάλντεν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως και το ελεγκτικό συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων και ο διαμεσολαβητής ελέγχει το έργο άλλων και προσπαθεί ε, να ενθαρρύνει τις καλύτερες πρακτικές οπότε λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη ε, το έργο της Επιτροπής των, Αρχών Ελέγχου Προπολογισμού που κάνουν ό,τι μπορούν για να εφαρμόσουν τις αρχές που θέλουμε να ενθαρρύνουμε άλλους να θετήσουν. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να γίνονται αποδεκτά τα σφάλματα, να αναγνωρίζονται όταν γίνονται και διορθώνονται και να υπάρξει σαν στόχος η συνεχής βελτίωσης ε, τούτων λεχθέντων. Χαίρομαι όλος ιδιαίτερος διότι δεν υπήρξαν ειδικέ παρατηρήσεις του ελεκτικού συνεδρίου ε, φέτος που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και να διορθώσουμε όμως πάντα ε, εξετάζουμε τι λέγεται για άλλα θεσμικά όργανα, κυρίως μικρά, μικρό θεσμικά όργανα για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ε, αντλήσουμε κάποια παραδείγματα και μαθήματα όσον αφορά τη συνεχή βελτίωση αν επιτρέπετε, Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ε, προσελκύσω την προσοχή σε δύο σημεία τα οποία επεξεργαζόμαστε. Πρώτα απ' όλα εσωτερική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών μας που έχει σαν στόχο αυτή ε, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα όσον αφορά την χρήση των ανθρωπίνων πόρων. Δεύτερον, αναλάβαμε την πρωτοβουλία να διαθέτουμε δημοσίες στην ιστοσελίδα του Δημοσιολογητού ε, το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και την, έκθεση, την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για να αυξηθεί η διαφάνεια ε, της διαχείρισής μας ε, και να γνωστοποιείται στο κοινό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χαδέ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Ντόξη του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εποπτείας ε, της ε, Προστασίας των Δεδομένων. Ευχαριστώ λοιπόν. Η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή Προστασία των Δεδομένων είναι μικρότερος και ο νεότερος φορέας στην οικογένεια των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Ο φορέας, όπως υπενθυμίστηκε ήδη, είναι ανεξάρτητη εποπτική αρχή από τη και το Εκτικό Συνέδριο και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα για την προστασία τη ιδιωτική ζωή και των προσωπικών δεδομένων γίνονται σεβαστά από τα θεσμικά όργανα και φορεί τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Επίση και όταν γίνεται, θεσπίζεται κάποια νομοθεσία. Είμαστε το μέσο στρατηγική μετριοπαθού αλλά συνεχού ε, μετρία αλλά συνεχού αναπτύξεω από την περίοδο 2007 μέχρι το 2013 και αυτή η στρατηγική ευθυγραμμίζεται με την πραγματική ανάπτυξη, αύξηση μάλλον του φόρτου εργασίας κατά αντίστοιχη περίοδο. Τα μέλη της Επιτροπής θα με καταλαβαίνουν όταν λέω ότι η δουλειά μας αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω του αντιχτύπου της συνθήκης της Λισαβόνας, διότι καινούργιοι τομεί έπρεπε να υποπτεύονται τεχνολογικές εξελίξεις όπως ε, η ψηφιακή ε, ατζέντα, μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στον αφορά την προστασία των δεδομένων και αύξηση της έμφασης που δίνει ο οργανισμός μας για την συμμόρφωση των θεσμικών οργάνων ε, και διαφόρων υπηρεσιών με αυτές τις αρχές που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Ευχαριστούμε το Κοινοβούλιο για την υποστήριξή του και βάσει υποστηρίξεως αυξήσαμε τα τελευταία τρία χρόνια τον προγραμματισμό μας και έχουμε πάει από, στο προσωπικό από 39 στους 43. 43 μέλη προσωπικού. Και αυτή η αύξηση του προσωπικού επετεύχθη με ταυτόχρονη μείωση του προϋπολογισμού διότι όπως και οι άλλοι φορείς ξέρουμε ότι χρειάζεται να κάνουμε οικονομίες. Οπότε ο προπολογισμό από 7,9 εκατομμύρια ευρώ το 2010 πήγε στα 7,6 εκατομμύρια ευρώ το 2012. Ε, ξεκινήσαμε μια διαδικασία εσωτερικών βελτιώσεων. Ξεκίνησαν αυτές το 2009, έγινε εσωτερική αναδιοργάνωση του φορέα τον Μάιο του 2010 και θα ήθελα να πω ότι μπορεί να δείτε τους καρπούς των προσπαθειών μας στη συνεχή βελτίωση της εκτελέσεως του προϋπολογισμού. Το 2009 είμαστε στο 73%, το 2011 στο 85% και προτιθέμεθα να πετύχουμε περαιτέρω βελτιώσεις. Και ξεκινήσαμε τώρα μια διαδικασία στατηγικής αναθεωρήσεως ε, φέτος και του χρόνου έγιναν εσωτερικές διαβουλεύσεις και αυτοαξιολόγησης ε, πέρσι και πρόκειται να ξεκινήσουμε και εξωτερική διαβούλευση ε, μαζί με τους εμπλεκομένους φέτος και θέλουμε να βελτιώσουμε τις, τον αντίκτυπο της προστασίας των δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των εργασιών μας. Επόμενο βήμα, το οποίο σχεδιάζουμε σε πλαίσια της αναθεωρήσεως, είναι να αναπτύξουμε βασικούς δείκτες επιδόσεων. Αυτό ήταν συγκεκριμένη ε, ε, σύσταση του Δ. Αγκαλέα του Ελεκτικού Συνεδρίου και να αναπτύξουμε και κάποιους εσωτερικούς δείκτες συνεχών επιδόσεων για να μπορούμε να προσμετρήσουμε τη βελτίωση των επιδόσεών μας και για πρώτη φορά, ίσως θα πείτε ώρα ήταν, αναπτύσσουμε ετήσιο και ενδιάμεσο ε, στατηγικό σχεδιασμό, οπότε θα έχουμε ετήσιο διαχειριστικό πρόγραμμα φέτος για πρώτη φορά και ενδιάμεσο στρατηγικό σχέδιο προγραμματισμού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Τόξη. Ευχαριστώ κύριε Τόξη. Οπότε ολοκληρώνουμε τις τοποθετήσει των εκπροσώπων των διαφόρων θεσμικών οργάνων και θα ήθελα να έχω κατά νου την ερώτηση που έδωσε ο κύριος Westlake. Δεν ξέρω κάποιος μπορεί να απαντήσει πώς μπορεί να νυχτερεύσει κανένας με 34 ευρώ. Μου φάνηκε ότι ήταν σημαντικό το θέμα αυτό, ίσως μια ηρωνική παρατήρηση. Υπάρχουν και άλλα θέματα βέβαια που είναι πολύ πιο σημαντικές στον αφορά τον ε, προπολογισμό. Καταρχήν θα ήθελα όμως να δώσω πάλι το λόγο στην κυρία Γιάλα Σέντρα, την εισηγήτριά μας. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. θα ακολουθήσω την ε, υπόδειξή σας. Ε, θα προσπαθήσω να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις στους υπεύθυνους από τα διάφορα θεσμικά όργανα και θέλω να ευχαριστήσω, επαναλαμβάνω, όλους που ήρθαν εδώ και για τις πληροφορίες που μας έδωσαν. Σε σχέση με το δικαστήριο, όπως πολύ καλά μας είπε ο εκπρόσωπος, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση Βέβαια αυτό δείχνει και ότι και οι πολίτες μπορούν να, να προσφύγουν στη δικαιοσύνη πλέον. Είναι θετικό δηλαδή από τη μία αυτό, ε, αλλά είναι και ανησυχητικό το ότι υπάρχει αυτή τόσο μεγάλη αύξηση των υποθέσεων. Το θετικό πάντως που συγκρατώ είναι ότι έχουν μειωθεί οι προθεσμίες. Βέβαια θα θέλαμε και μεγαλύτερη μείωση εμείς, αλλά σε σχέση με άλλα δικαιοδοτικά όργανα, με άλλα δικαστήρια εθνικά, είναι κάτι που πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα το δικαστήριο να ρωτήσω, πώς, με ποιο τρόπο χρησιμοποιείται το σύστημα το οποίο ονομάζεται κούρια, το ε, ηλεκτρονικό δηλαδή αυτό εργαλείο, πώς μπορείτε να βελτιώσετε την διαχείριση και λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των ε, υποθέσεων, πώς θα βελτιώσει τις προθεσμίες και τη διαχείριση των υποθέσεων. Προς το ελληνικό συνέδριο, καταρχάς ε, θέλουμε να ευχαριστήσουμε το ελεκτικό συνέδριο τη βοήθειά του, αλλά έχουμε απαιτήσει. Ε, συνεχίζουμε να θέλουμε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, καλύτερη διαχείριση, αλλά σίγουρα να γνωρίζουμε τι προσπάθειε που έχει καταβάλει το ελεκτικό συνέδριο. Ένα ερώτημα. Πολύ συγκεκριμένο. σε σχέση με αυτά που είπε και ο εκπρόσωπος δηλαδή ότι θα ξεκινήσει το λεγόμενο peer review, δηλαδή αναθεώρηση από ομοτήμους. Συγκεκριμένα, ποιες είναι οι προθεσμίες, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και κάτι που ζητάμε και διεκδικούμε ανέκαθεν να υπάρχει κάποια δημοσιοποίηση ε, των ε, στοιχείων από το ελεγκτικό συνέδριο για τις θέσεις και όχι να τα κρατούμε έτσι μυστικά όλα αυτά. Για το επόμενο θεσμικό όργανο κάτι πολύ γενικά σε, ε, στο συντονισμό. Για ε, τον κύριο Γουέσλη συγκεκριμένα θέλω να θέσω το ερώτημα. Πώς αξιολογείται από την Επιτροπή των Περιφερειών τις προσπάθειες διοικητικής συνεργασίας, που είναι και ένα παράδειγμα καλής ε, συνεργασίας και διαχείρισης. Προς την ΕΟΚΕ τώρα, την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή, να αναγνωρίζω την προσπάθεια που έχουν καταβάλει τα μέλη της για να ικανοποιήσουν ένα πάγιο αίτημα του Κοινοβουλίου να υπάρχει ένα καταστατικό, ένα καθεστώς ε, συμβούλου που έχει να κάνει με την αποζημίωση των εξόδων μετακίνησης, ε, την ημερήσια αποζημίωση κτλ. 34 ευρώ ίσως να σας φαίνεται ε, κάτι απίθανο, όμως όλα μπορούν να συμβούν κύριε Πρόεδρε. Και από ό,τι μα είπαν, δεν είναι η μόνη μερική αποζημίωση, υπάρχει και άλλη μια αποζημίωση για την προετοιμασία των εργασιών των συνόδων. Θα ήθελα λοιπόν να μα πει εκπρόσωπο τη ΕΟΚΕ πώ αθρίζονται και πώ αλληλοεπικαλύπτονται, αν θέλετε, οι αποζημιώσει του άρθρου 11 και του άρθρου 12 σε σχέση και με τα έξοδα μετακίνηση και την επιστροφή των εξόδων αυτών. Έχουμε ζητήσει να υπάρχει διαφάνεια εμεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να μα ε, ε, πει ο Γενικό Γραμματέα τι άποψη έχει για ένα έντυπο. Τι είδου έντυπο είναι αυτό που φαίνεται εκεί αν έχουν παραστήσει συνεδριάσεις ε, οι σύμβουλοι και τι γίνεται με τα έξοδα μετακίνησης. Και σε ό,τι αφορά τη βιντεοδιάσκεψη είναι λίγο περίεργο. Ναι, μεν μιλάμε για έξοδα μετακίνησης, για συμμετοχή σε βίντεο διασκέψεις, Ίσως αυτό να σημαίνει ότι από το χωριό τους πηγαίνουν σε μια πόλη οι σύμβουλοι. Αλλά μας φαίνεται λίγο περίεργο να παίρνουν να έχουν μια επιστροφή εξόδων μετακίνησης για να συμμετάσχουν σε βιντεοδιασκέψεις. Θα ήθελα να μας το εξηγήσει αυτό ο Γενικός Γραμματέας. Και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ΕΟΚΕ, θα ήθελα να μας εξηγήσει ο εκπρόσωπος τι γίνεται με την υπόθεση που διερευνάει όλα αυτή τη στιγμή είχαμε και δύο παρεμβάσεις του διαμεσολαβητή σχετικά. Και το δικαστήριο της δημόσιας διοίκησης ε, έχει επιληφθεί αυτή τη υπόθεση. Είναι ένα θέμα που μας ανησυχεί και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Υπάρχει περίπτωση whistleblowing και ο συγκεκριμένο ε, μάλλον θα αντιμετωπίσει και κάποια προβλήματα. Ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα. Θα θέλαμε να μα εξηγήσετε. Και τι έγινε και με την ε, ε, προκήρυξη της θέσης του που υπήρχαν κάποια σφάλματα στη διαδικασία. και δεν, έγιναν, δεν τηρήθηκαν οι όλες προθέσεις και τα χρονοδιαγράμματα όπως θα έπρεπε. Σε ό,τι αφορά το διαμεσολαβητή, τον Νόμουτσμαν, φυσικά και συμφωνούμε ότι έχει ως στόχο τον εξορθολογισμό της διαχείρισης, βελτιώνεται κάθε μέρα η διαχείριση, το βλέπουμε, αλλά Αυξάνονται οι καταγγελίες των οποίων επιλαμβάνει το διαμεσολαβητής. Με ποιο τρόπο καταφέρνει ή έχει καταφέρει να μειώσει τις προθεσμίες. Και τι γίνεται με τη διαχείριση, τηλεματική, νέες τεχνολογίες, πώς μπορεί να αξιοποιηθούν όλα τα εργαλεία αυτά για να μειωθούν ακριβώς οι προθεσμίες απάντησης. Το Κοινοβούλιο είχε εκπονήσει και ειδική έκθεση για το διαμεσολαβητή. Αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση και σε ό,τι αφορά τον επόπτη δεδομένων που τον καλωσορίζουμε γιατί έχουμε επιτέλους στοιχεία στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να εργαστούμε σε βάθος και σε σχέση με την απαλλαγή. Σας ευχαριστούμε για τον εξορθολογισμό και τις προσπάθειες που καταβάλλετε. Αλλά έχουμε και ένα ερώτημα. Συγκεκριμένα, πώς διορθώνονται, πώς προσπαθείτε να διορθώσετε τα σφάλματα τα οποία παρατηρήθηκαν στις διάφορες εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Ιδίω σε σχέση με την ΤΑΣ ε, του 2009, την ε, πρώτη ΤΑΣ του 2009. Σίγουρα, εντάξει, τώρα ξεκινάτε, το καταλαβαίνουμε, αλλά πώς μπορούν να διορθωθούν αυτά τα σφάλματα και σε ό,τι αφορά ε, την ε, λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος ε, που δρομολογήθηκε, μιλάμε για ευαίσθητα δεδομένα, το καταλαβαίνουμε αυτό. Πώς μπορείτε λοιπόν να εξασφαλίσετε, να κάνετε πιο ασφαλή τη διαχείριση των διαφόρων φακέλων και αρχείων. Τώρα, στο σχέδιο δράσης και στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων, για το 2011 μιλάω ήδη, μπορέσατε να καταρτήσετε κάποιους δείκτες αποτελεσματικότητας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση προβλέπετε επίσης να έχετε ένα κεφάλαιο στην αιτήσια έκθεση πεπραγμένων, το οποίο θα είναι αφιερωμένο στην παρακολούθηση των προτάσεων ψηφίσματος για την απαλλαγή. Ουσιαστικά αυτά είχα να πω. Και βέβαια θα ακούσουμε και τα ερωτήματα που θα έχουν και οι συναδελφοί μου. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Συγγήτρια. Ε, για το ΕΛΚ ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Dann Frau Ivanova, vielleicht. Thank you, Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους των διαφόρων ε, θεσμικών οργάνων για τις παρεμβάσεις τους. Στο ψήφισμά μας για την απαλλαγή το 2009 για την Επιτροπή των Περιφερειών ζητήσαμε αναθεώρηση όλων των τομέων των δαπανών για να εντοπιστούν ε, τυχόν οικονομίες. Και έχω ερώτημα προς όλους τους εκπροσώπους. Μπορείτε να μας πείτε κατά πόσο αυτή η αναθεώρηση έλαβε χώρα στον οργανισμό σας και αν ναι, ε, τι δράσεις ανελήφθησαν σχετικά με αυτό, διότι νομίζω ότι σε εποχές λιτότητας είναι σημαντικό κάθε φορέας να καταβάλει προσπάθεια για βελτιστοποίηση των δαπανών. Και άλλο ερώτημα αφορά ειδικά την εποπτική αρχή για την προστασία των δεδομένων η κυρία Συγήτρια, η κυρία Γιάλα, ρώτησε ποια είναι η γενική συνέχεια που δόθηκε στη στάση του ελεκτικού συνεδρίου, αλλά εγώ θέλω συγκεκριμένο ερώτημα όσον αφορά την εξ των υστέρων μηχανισμό επαλήθευσης, συγκεκριμένη σύσταση του ελεκτικού συνεδρίου που δεν εφαρμόστηκε Κάνατε κάτι πάνω σε αυτό. Τι πρόοδο σημειώσατε, διότι είναι πολύ σημαντικός εκ των υστέρων έλεγχος για την ε, βελτίωση των ε, συστημάτων ελέγχου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πένοβα. Ο κύριος Βόρκιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προς τον κύριο Βέστλινγκ. έχω το ερώτημα από την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή όχι για τα 34 ευρώ, αλλά για την ε, οικονομική διαχείριση. Αν τα καταφέρουν συνάδελφοι με 34 ευρώ την ημέρα, σίγουρα ε, χειρίζονται πολύ καλά τα οικονομικά. Ε, ερώτηση. Ε, όσον αφορά την απαλλαγή του 2009 και ανησυχίε που εκφράστηκαν. Κύριε Βέσλεϊ, ποιε αλλαγέ πρέπει να γίνουν. Ποιε έγιναν από το 2009, μάλλον. Ποιε αλλαγέ. Αναφέρθηκε στα διπορικά και άλλες αποζημιώσεις. Έχουμε άλλα παραδείγματα λαγών. Θεωρεί ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω βελτιώσεων. Προπολογισμό 2010. Ερώτηση. Εξέφρασε ανησυχίε στο ελεκτικό συνέδριο προ τον κύριο Βέσλικ ή θεωρεί ότι η Επιτροπή έχει κάνει πρόοδο πραγματική όσον αφορά την οικονομική διαχείριση. Τρίτη ερώτηση. Τι μέτρα διαφύλαξης υπάρχουν τώρα, ούτω ώστε οι αποφάσεις τα οικονομικά και τους πόρους ε, τεκμηριώνονται και δικαιολογούνται σωστά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έπινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εποχέ λιτότητα περνάμε. Το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο κάνουν προσπάθειε για περικοπέ. Και οι προπολογισμοί τη ΟΚΕ και τη Επιτροπή των Περιφερειών εξακολουθούν να αυξάνονται. Περίπου 50% την τελευταία οκταετία. Άρα, περιορισμένοι πόροι, αυτή η διατύπωση που ανέφερε ο κ. Βέστλικ ε, και ο κ. Στάλ είναι μάλλον ε, πολύ μετριοπαθής διατύπωση. Σε ένα χρόνο η ΟΚΕ και η Επιτροπή των Περιφερειών αύξησαν κατά 1,5% στους υπολογισμού και 2,9% αντίστοιχα στα 130 εκατομμύρια για την ΟΚΕ και 86,5 εκατομμύρια ευρώ για την Επιτροπή των Περιφερειών. Υπάρχει κάτι που είναι σημαντικό βέβαια. Το ψήφισμα της 10ης Μαΐου του 2011 και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την ΟΚΕ να εφαρμόσει μια γενική αναθεώρηση των δαπανών όλων των τομέων δραστηριοτήτων, ούτω ώστε πράγματι να αποδίδουν τα χρήματα που δαπανώνται. Εντύπωσή μου, Πρόεδρε, είναι ότι η Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή ε, τελικά προσπαθεί να αποφύγει τον έλεγχο. Κινείται κάτω το επίπεδο του ραντάρ, με λόγια. Και, πότε θα η μελέτη, δημοσιοποιηθεί, με ενδιαφέρει. Το ελεκτικό συνέδριο αναφέρθηκε στο σύστημα επιστροφών, δαπανών, όπου η ΟΚΕ, τα μέλη της ΟΚΕ παίρνουν κατά αποκοπήν ποσά κατά συνεδρίαση χωρίς να αποδεικνύουν τις δαπάνες. Σε άλλα θεσμικά όργανα έχουν κατασταθεί αποκοπήν, κατά αποκοπήν ε, πληρωμές και ζητείται απόδειξη για να κατευθύνουν αποζημιώσεις. Συνεχίζει μέχρι το 2015 αυτό το σύστημα η ΟΚΕ. Γιατί δεν το καταργεί αμέσως. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Ιστορικά, όπως γνωρίζουμε, το σύστημα κατά αποκοπήν ε, υπήρξε αντικείμενο μεγάλων καταχρήσεων. Όπως ο κ. Τζάκο Μοριγκάλτο της ΟΚΕ επήρε, ε, καταδικάστηκε φυλάκη, σε φυλάκιση με αναστολή διότι πήρε από διάφορες φορείς της Ιταλίας εκπροσώπους ε, εργοδοτών χρήματα και από την ΟΚΕ. Ούτε πρόστιμο πλήρωσε, ούτε τις ε, αχρεωστήτως καταβληθήσεις αποζημιώσεις. Μιλάμε για εισρωή χρημάτων. Πρέπει να μιλάμε και για εκροές χρημάτων. Και οι δύο επιτροπές λένε ότι συμμετέχουν σημαντικά στη συμμετοχική δημοκρατία. Δεν υπάρχει απόδειξη όμως γι' αυτό, μεγάλες αποδείξεις, παρόλο που εκεί τριπλασίασε τον προπολογισμό για επικοινωνία την τελευταία τριετία. Η Επιτροπή των Περιφερειών σχεδόν διπλασίασε τα ανάλογα κονδύλια. Όσον αφορά 0,35% των συνολικών επισκεπτών ε, στον ιστοσελίδα europa.eu για την Επιτροπή των Περιφερειών είναι 0,27% το ποσοστό επισκεπτών. Ε, δεν χρησιμοποιούν καθόλου καλά τα κοινωνικά μέσα που είναι πηγή αλλαγών στον κόσμο. Είναι επανάσταση. Και οι δύο επιτροπές έχουν λιγότερα like στο facebook ή twitter από ό,τι έχουν προσωπικό. Και η Επιτροπή των Περιφερειών δεν έχει ανακαλύψει τον, ε, το Twitter. Ο κύριος Στάλ δεν υπάρχει στο Twitter. Κύριε Πρόεδρε, τι έγινε το ψήφισμά μας το Μαΐου 2011 για την απαλλαγή του προπολογισμού 2009. Τι δείχνει η μελέτη. Καμία από τις δύο επιτροπές δεν κάνουν αυτά που σχέθηκαν και προσπαθούν να αποφύγουν περικοπές δαπανών. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε πόσο είναι χρήσιμε οι επιτροπέ εδώ. Το 2003, πρώην συνάδελφο, η κυρία Χέλα Τόνεν Σμιτ, υπέβαλε μια εργασία στην συνέλευση για τη συνταγματική συνθήκη και είπε ότι okay, και είπε δεν είναι εστιασμένη, πολύ δαπανερή, πολύ αναποτελεσματική. Η κυρία Χέλα Τόνεν Σμιτ είναι πρωθυπουργό τη Δανία και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως του Συμβουλίου, προεδρεύουσα. Θα πρέπει να μην δώσουμε την απαλλαγή στην ΟΚΕ και στην Επιτροπή των Περιφερειών εάν δεν κάνουν σοβαρές προτάσεις για περικοπή ε, των δαπανών. Και πρέπει να καλέψουμε και τους δύο γενικούς γραμματείς εδώ και να ακούσουμε τι έχουν να προτείνουν για να ευθυγραμμιστούν με το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δύο και τη μελέτη που είχα αναθέσει να γίνει θα τη διαθέσω και σε εσά κύριε Πρόεδρε και στα μέλη τη Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Έπινγκ. Κάτι έμαθα λοιπόν. Ε, ε, είμαστε στο διαδίκτυο. Είναι ενδιαφέρον. κάποιο θα μπει στο Twitter και αναρωτιέμαι τι κάνει ο κόσμος εδώ γύρω με τα κομπιούτερ. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ζητήσουμε τώρα του εκπροσώπου των ε, φορέων αυτών κατά πόσο μπαίνουν στο Twitter ή όχι. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να συνδυαστεί με το ελεκτικό συνέδριο. Άλλος της θέλει να υποβάλει ερώτηση ή μπορούμε να περάσουμε στις απαντήσεις. Η κυρία Γκέσλα. Λοιπόν, προσπάθησα να δω πόσους έχουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπαλλήλους γενικά. Όποιο το προσπαθήσει αυτό έχει πολλή δουλειά να κάνει γιατί δεν υπάρχει ένα έγγραφο έτοιμο. Θα πρέπει κανένα να κάνει του υπολογισμούς μόνο του. Έχουμε μόνιμους υπαλλήλου, επισυμβάσει, προσωρινού, Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όλα τα θεσμικά όργανα να μας δώσουν τις πληροφορίες αυτές για το έτος 2011. Όλων των ειδών τους ε, εργαζόμενους να περιλάβουν στους καταλόγους αυτούς πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα να υπάρχει ένα τέτοιο έγγραφο έτοιμο χωρίς να πρέπει κανένας να ασχολείται ε, με τις ώρες. Γιατί νομίζω ότι είναι πολύ δυσάρεστο να μην ξέρει κανένας πόσους υπαλλήλους έχουμε γενικά και εργαζόμενους. Περίπου 55.000 είναι αν σας ενδιαφέρει. Αλλά θα ήθελα να το ξέρω με μεγαλύτερη ακρίβεια και γι' αυτό παρακαλώ τους παρόντες να σκεφτούν πώς μπορούν να ενώσουν τα στοιχεία αυτά και να μας τα δώσουν για να ξέρουμε πού μπορούμε να τα βρούμε αν τα χρειαζόμαστε κάπου. Πρόεδρος, ναι, πολύ σημαντικό το σημείο αυτό. Δεν υπάρχει λοιπόν φαίνεται παγιωμένη βάση στοιχείων. Για να είναι συγκρίσιμα θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη ημερομηνία νομίζω. Τέλος πάντων, άλλος που θα ήθελα το λόγο δεν έχει ζητήσει κανείς. Θα ήθελα λοιπόν να περάσω στη σειρά Όπω είχαν προηγουμένω για να δοθεί μια απαντήση. Ο κ. Καρότς πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για την ερώτηση σε σχέση με το σύστημα κούρια, Ένα σύστημα το οποίο μπορούν να, να ε, χρησιμοποιήσουν οι διάδικοι για να στείλουν ε, τα δικόγραφα στο δικαστήριο. Και τα τρία επίσης δικαστήρια μπορούν μέσω αυτού του συστήματος να κοινοποιήσουν κάποια έγγραφα. Δεν χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή το Twitter για να επικοινωνούμε με τους διαδίκους, αλλά το σύστημα e-Courier είναι ένα σύστημα πληροφορικής, το οποίο το δικαστήριο ε, μετά από προετοιμασία μακρά ε, και σε πλήρη συνεργασία πρέπει να πω με τις υπηρεσίες πληροφορικής της Κομισιόν, πάρα πολύ καλό παράδειγμα διοργανικής συνεργασίας, ε, το δρομολόγησε λοιπόν ε, την 1η ε, Νοεμβρίου 2011 αυτό το σύστημα και πρέπει να πω με πολλή επιτυχία. Οι διάδικοι ε, μας λένε ότι είναι ένα σύστημα το οποίο διευκολύνει τα διοικητικά καθήκοντα γιατί πρέπει να σταλούν σε πολλαπλά αντίγραφα, τα διάφορα έγγραφα <clears throat> και να είναι και πιστοποιημένα. Μειώνεται το κόστος και για το δικαστήριο είναι πολύ σημαντικό κομμάτι η μηχανοργάνωση των εσωτερικών εργασιών. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ηλεκτρονική επεξεργασία των υποθέσεων. Βέβαια δεν σημαίνει ότι απλουστεύεται η επίλυση των υποθέσεων επειδή στέλνονται ηλεκτρονικά κάποια έγγραφα, αλλά σίγουρα επιταχύνονται ε, οι διαδικασίες τουλάχιστον λήψης της τεκμηρίωσης. Αυτό είναι σημαντικό και αυτό κατατείνει προς τον εξυγχρονισμό ε, του δικαστηρίου. Βέβαια υπάρχουν ταυτόχρονα και πολύ σημαντικές οικονομίες που γίνονται, εξοικονομήσεις πόρων. Εμείς ε, βλέπουμε σε κάθε περίπτωση ως δικαστήριο που μπορούμε να εξοικονομήσουμε πόρους, χωρίς να υπονομεύσουμε βέβαια και την ποιότητα του νομικού και δικαστικού μας έργου και πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή προσανατολιζόμαστε προς ε, εγκατάλειψη ε, της ε, δημοσίευσης σε έντυπη μορφή των ανθολογιών της νομολογίας και θα τις δημοσιεύουμε τις υποθέσεις ηλεκτρονικά, την ομολογία δηλαδή, και αυτό σίγουρα θα ε, έχει ως αποτέλεσμα πολύ σημαντική, σημαντικές οικονομίες, αλλά και ο πολίτης που ενδιαφέρεται για τη δικαστική δραστηριότητα θα μπορεί να ενημερώνεται καλύτερα. Είμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή σε, ε, αυτή τη διαδικασία της ε, μείωσης λοιπόν του κόστου, τη βελτίωση λειτουργίας του οργάνου μας με αυτή την ηλεκτρονική δημοσίευση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καλότ. Για το ελεκτικό συνέδριο ο κύριος Ζωής Καρσία έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση με το πρώτο ερώτημα, το οποίο είχε να κάνει με το peer review, την αναθεώρηση εξ όλες Πρέπει να σας πω ότι το ελεγκτικό συνέδριο έχει ήδη ξεκινήσει τη σχετική προετοιμασία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση της επιλογής των ελεγκτικών συνεδρίων που θα μπορούσαν να κάνουν αυτή την αναθεώρηση, αυτή την αξιολόγηση. Και θα του στείλουμε τη σχετική εντολή. Την αναθεώρηση θα ε, την ε, δημοσιεύσουμε στη διάρκεια της, ε, τρέχουσα, της χρονιάς αυτής. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι τον κώδικα διοντολογίας τον επεξεργαζόμαστε, τον αναθεωρούμε. Μιλάω για τον κώδικα διοντολογίας του προσωπικού. Έχει γίνει αυτό άλλωστε και από άλλα θεσμικά όργανα και τις επόμενες εβδομάδε πιστεύω ότι θα μπορούσα να σας δώσω μια θετική απάντηση στο ερώτημά σας κυρία Επίσης, ό,τι αφορά την ώρα της κυρίας Γκρέσλε, στην περίπτωση του ελεγκτικού συνεδρίου, τον Ιανουάριο, τα τέλη συγκεκριμένα του 2011, είχαμε 887 ε, υπαλλήλους, 58 συμβασιούχους, 11 εθνικούς εμπειρογνώμονες και 17 υποτρόφους εκπαιδευόμενους συνολικά 973 άτομα προσωπικό. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε για το 2011. 2010-2011 και θα όλα τα στοιχεία τα διαβιβάσουμε στην εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ρουίς Καρσιά. Ε, είναι καλό να τα μαζέψουμε τα στοιχεία αυτά νομίζω και κάποια συγκεκριμένα ημερομηνία. Μετά θα δώσω το λόγο στο Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής των Περιφερειών, τον κύριο Στάλ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Όσον αφορά τι ερωτήσει που επιβλήθησαν, έχω να πω τα εξή. Καταρχήν, σε ερωτήσει τη εισηγήτρια, όσον αφορά την συνεργασία με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Για την Επιτροπή των Περιφερειών έχουμε τους περισσότερους ε, απασχολούμενους στις κοινέ υπηρεσίες. Υπηρεσίες δηλαδή από κοινού με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή που έχουν οργανωθεί για να δράσουν αποτελεσματικά παραδείγματο χάρη τα κτίρια, τα μοιραζόμαστε, τις υπηρεσίε μετάφραση, το κειμένο μοιραζόμαστε γιατί αυτά όλα οδηγούν σε εξοικονομήσεις μεν αλλά και σε συμπληρωματικά προβλήματα συντονισμού. Υπάρχει μια ε, συνθήκη συνεργασίας που μας δίνει τη δυνατότητα να λύσουμε τα προβλήματα αυτά. Έχουμε νομίζω τώρα και καλό πολιτικό έλεγχο της διαχείρισης και γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή η συνεργασία των δύο θεσμικών οργάνων για τις περισσότερες διοικητικές τους διαδικασίες είναι καλό παράδειγμα για εξοικονομήσεις που μπορούν να γίνουν και περαιτέρω σε συνεργασία τα οργάνων. Γιατί κάτι τέτοιο μπορεί οπωσδήποτε να οδηγήσει σε εξοικονομήσεις. Θα ήθελα επίσης να συμπληρώσω το θέμα της δήλωσης των ε, οικονομικών συμφερόντων των μελών μας. Είναι ένα θέμα που έχει θίξει το Κοινοβούλιο τα μέλη της μας ε, ακολουθούν, ε, εκπληρούν αυτές τις επιθυμίες του Ευρωπαϊκού, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή σε τακτά χρονικά διαστήματα υποβάλλουν δήλωση όσον αφορά την οικονομική τους κατάσταση και ο πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών αποφάσισε οι δηλώσεις αυτές να δημοσιεύονται στη ισοσελίδα της Επιτροπής μας για να μπορέσουμε έτσι να πληρώσουμε τις επιθυμίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να είναι γενικά διαθέσιμα τα στοιχεία αυτά. Όσον αφορά τώρα τις εξοικονομήσεις. Αυτό είναι κάτι οπωσδήποτε σημαντικό σε, περίπτωση, σε περίοδους κρίσης και για τα μέλη μας που είναι ε, εκπρόσωποι τοπικών ομάδων, δήμαρχοι κλπ. Είναι όλοι άτομα που πλήττουν ιδιαίτερα από τις εξονομήσεις που οφειλούν στην κρίση και γι' αυτό απαιτούν το Ευρωπαϊκό Όργανο στο οποίο ενεργάζονται να υιοθετήσει επίσης κάθε απαραίτητο μέτρο για να γίνουν εξοικονομήσεις. Και γι' αυτό θα ήθελα πάλι να τονίσω ότι η Επιτροπή των Περιφερειών έχει υποβάλει ένα πρόγραμμα για τη βελτίωση της διοικητικής μεταρρύθμισης και να οδηγηθεί έτσι σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Έχουμε 54 μέτρα υποβάλει για τη βελτίωση της διοίκησης. Και το Προεδρείο παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα την εξέλιξη με τα μέτρα αυτά. Εξετάσαμε όλα τα κονδύλια του προπολογισμού μας εν ώψη των συζητήσεων για τον προπολογισμό και κάναμε περικοπές όπου μπορούσαμε. Εκεί που είναι δύσκολο βέβαια είναι να περικόψουμε στις πολιτικές δραστηριότητες, γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, η Επιτροπή των Περιφερειών μέσα στα πλαίσια των αλλαγών που επέφερε η συνθήκη της Λισαβόνης απέκτησε νέες αρμοδιότητες, τις οποίες πρέπει να πληρούμε. Θα ήθελα ταυτόχρονα όμως να αναφέρω ότι ακριβώς ενώπιση των εξοικονομήσεων ήταν δυνατό στον τομέα των κτηρίων να πετύχουμε το πιστοποιητικό εμάς για τα κτίρια, για την πολιτική μας για τα κτίρια. Και έτσι μπορέσαμε να κάνουμε σημαντικές ε, εξοικονομήσεις όσον αφορά την ενέργεια για το φυσικό αέριο παραδείγματος κάνει της άξου 30%. Προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε κατανοητών αποτελεσματικοί. Όσον αφορά τώρα το θέμα της ε, ε, επίδραση της Επιτροπής των ε, Περιφερειών και το ανέφερε νομίζω πολύ καλά ο κύριος Έπινγκ. Είναι ένα θέμα που συζητάμε και μεταξύ των μελών μας. Σύμφωνα με τον κανονισμό μας έχουμε την υποχρέωση μία φορά το χρόνο να υποβάλουμε μία έκθεση για την αποτελεσματικότητα των εργασιών μας. να πούμε δηλαδή κατά πόσον ο χρόνος που διαθέτουν οι πολιτικοί αυτοί που έχουν έργο να επιτελέσουν στη χώρα τους, κατά πόσον λέω αυτός ο χρόνος που δαπανήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δαπανήθηκε σωστά, αξιόλογα. Αυτό το θέμα δηλαδή των επιπτώσεων ενός θεσμικού οργάνου είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα και αυτό έχει πιο σημαντικά ερωτήματα που θα πρέπει να θέτουν σε αυτούς οι ίδιοι πολιτικοί. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιο είναι το επίκεντρο των εργασιών μας. Ε, εμείς δεν έχουμε σαν στόχο να έρθουμε σε άμεση επαφή με κάθε ένα πολίτη. Και γι' αυτό το θέμα του Twitter είναι βέβαια ενδιαφέρον, αλλά η ο δική μας ομάδα στόχος είναι οι 90.000 τοπικές ομάδες και οργανισμοί. Οι δήμαρχοι, οι τοπικοί υπουργοί, η τοπική αυτοδιοίκηση, αυτή είναι η δική μας εταίροι. Και γι' αυτό έχουμε μια στενή συνεργασία και με τις διάφορες ενώσεις αυτών των οργανώσεων, όπου υπάρχουν διάφορα εφημερίδες, διάφορα ενημερωτικά δελτία, που έχουν σαν στόχο την επαφή με αυτή την ομάδα του πληθυσμού που προσωπούν οι δικοί μας, τα δικά μας μέλη δεν νομίζω ότι ε, μπορεί ένας μικρός οργανισμός σαν το δικό μας που έχει ένα προπολογισμό μικρότερο από πολλών δήμων και κοινοτήτων μπορεί να επικοινωνήσει λέω με κάθε ένα πολίτη. Εμείς επικοινωνούμε με τις ομάδες στόχο όσον αφορά τώρα τις ερωτήσεις της κυρίας Γκρέσλε. Ευχαριστώ να τη δώσουμε όλες τις πληροφορίες για το προσωπικό που έχουμε εμείς και που όπως σας είπα είναι πάρα πολύ λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Στάλ. Ο κύριος Westlake για την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μετά από όσα είπε ο συνάδελφος και αρχαριστάς για τις κοινέ υπηρεσίε. νομίζω κύριε Πρόεδρε εσείς ήσασταν αυτός που έθεσε το σχετικό ερώτημα, νομίζω ότι θα πρέπει τα άλλα θεσμικά όργανα να ε, μάθουν περισσότερα για την ε, συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των επιτροπών, τις κοινέ υπηρεσίες, διότι είναι ένα καλό παράδειγμα, ίσως και ένα μοντέλο για τη μελλοντική συνεργασία, αν θέλουμε να έχουμε οικονομίες η δική μας συνεργασία βασίζεται σε μια συμφωνία συνεργασίας. Είναι ετούς διάρκειας, είμαστε στη μέση και κάναμε και την διάμεση αξιολόγηση πέρυσι, η οποία ήταν άκρος θετική. Ο Γκέρχαρτ Στάλ και εγώ προσωπικά επιβλέπουμε ένα πολύπλοκο σύστημα διακυβέρνηση, το οποίο λειτουργεί όμω, διότι είμαστε αποφασισμένοι και οι δύο γι' αυτό. Και συγχρόνω εξοικονομούμε σημαντικού πόρου για τον Ευρωπαίο Φορολογούμενο και Ψηφοφόρο. Με τα χαρά να σας δώσουμε περισσότερε πληροφορίες για το πώ ε, λειτουργεί αυτό το σύστημα. Να σα πω όμω ότι είναι πολύ σημαντική μορφή συνεργασία. Για παράδειγμα, στην περίπτωση τη ΕΟΚΕ, σχεδόν πάνω από του μισού ανθρώπινους πόρου που έχουν βρίσκονται στι κοινέ υπηρεσίε. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτό το σύστημα. Εθέθησαν κάποια ερωτήματα. Αρχίζω από τα ερωτήματα τη ηγήτριας για το νέο χρηματοοικονομικό καθεστώ των μελών. Πρέπει να σα ομολογήσω ότι και εγώ δεν είχα επαρκή γνώση και αντίληψη της κατάστασης πριν ε, γίνω μέλος Επιτροπής για το πώς εργάζονται τα μέλη της Επιτροπής. Πρέπει να υπογραμμίσω ότι δεν λαμβάνουν ευρωπαϊκό μισθό, σε καμία περίπτωση. Τον μόνο μισθό τον οποίο λαμβάνουν είναι ο μισθός που λαμβάνουν από την οργάνωση που εκπροσωπούν. Επομένω, όταν ένα μέλος δεν είναι παρόν στην οργάνωση του ή της, γιατί ε, ασχολείται με το έργο της Επιτροπής μας, αντιπροσωπεύει ένα κόστος για την οργάνωση ε, που εκπροσωπεί. Σε πολλές περιπτώσεις, πολλά μέλη μας, ε, για πολλά μέλη μας το λαμβάνουν αυτό υπόψη οι οργανώσεις τους ό,τι αφορά τις αποδοχές τους. Αυτό δεν είναι παρκώς κατανοητό. Δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά τα μέλη της ΕΟΚΕ είναι ουσιαστικά Ευρωπαίοι θελοντές. Δεύτερο ερώτημα. Πόσος χρόνος απαιτείται για να ε, ασχοληθεί κάποιο με τι εργασίε τη Επιτροπή μα. Ένα Μαλτέζο για να έρθει ε, στι Βρυξέλλε ε, πρέπει να λείψει τουλάχιστον δύο-τρει μέρε από το γραφείο του στη χώρα του. Η βιντεοδιάσκεψη στο μέλλον, αν καταφέρουμε να επιλύσουμε κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά τη διερμηνία, ίσω να αποτελέσει ένα τμήμα τη λύση. Ένα μέλο όμω τη ΕΟΚΕ, εάν συμμετέχει σε μια βιντεοδιάσκεψη, δεν είναι στα γραφεία τη οργάνωσή του. Εξού και η λογική που διέπει αυτό το νέο χρηματοοικονομικό καθεστώ. Θα ήθελα να σας δώσω τις πληροφορίες ε, και συγκεκριμένα στην εισηγητρία θα τις διαβιβάσω και το σχέδιο απόφασης και οποιαδήποτε άλλη επεξήγηση ε, χρειαστεί. Υπήρξαν επίσης ερωτήματα για την Όλαφ και για το διαμεσολαβητή. Να πω ότι η ΕΟΚΕ πάντοτε, πάντοτε συνεργαζόταν και συνεργάζεται πλήρως με όλους αυτούς τους οργανισμούς ε, και θεσμικά όργανα, όπως ο διαμεσολαβητής ε, ή το ελεκτικό συνέδριο. Η κυρία Γιάλα, νομίζω πρώτα ρώτησε για την Όλαφ. Δεν νομίζω ότι θα σας αποκαλύψω κάποιο κρατικό μυστικό αν σας πω ότι η Όλαφ πράγματι δρομολόγησε στις 11 Μαρτίου του 2011 μία έρευνα. Εμείς συμμορφωθήκαμε πλήρως και συνεργαστήκαμε απόλυτα. Αφορούσε μια πειθαρχική διαδικασία η οποία είχε ξεκινήσει το 2005-2006 με την υποτιθέμενη κλοπή 250 ευρώ. Στην πειθαρχική διαδικασία τελικά δεν προέκυψε ότι ήταν βάσιμη αυτή η καταγγελία. Ε, δεν έχουμε ακούσει κάτι έκτοτε. Εμείς σίγουρα συμμορφωνόμαστε και θα συνεχίσουμε να συμμορφωνόμαστε με την Όλαφ και τις υποδείξεις της όταν ε, υπάρχει κάποια έρευνα στο μέλλον από πλευρά τη όλα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το διαμεσολαβητή. Και εμεί ε, προσπαθούμε να τηρήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο τι συστάσει του διαμεσολαβητή. Και νομίζω ότι μα ανέφερε στην περσινή του έκθεση ω καλό παράδειγμα ενό θεσμικού οργάνου που προσπαθεί πάντοτε να βρει φιλικού διακανονισμού και λύσει. Μία περίπτωση, μία υπόθεση υπάρχει, είναι αρκετά πολύπλοκη και χρονοτριβή, καθυστερή Είχαμε μιλήσει με το Διαμεσολαβητή το Δεκέμβριο και εγώ προσωπικά πήγα στις υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή την προηγούμενη εβδομάδα, στο Στρασβούργο δηλαδή, για να του δώσω περισσότερα στοιχεία σε σχέση με την υπόθεση. Ε, εγώ για ε, αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση έχω μάθει πιο πολλά από όσα θα ήθελα αν θέλετε να μάθω έχουν γίνει κάποιες εσωτερικές ε, μεταρρυθμίσεις στην Επιτροπή μας ό,τι αφορά τις διαδικασίες προαγωγών. Ελπίζω να βρούμε στο μέλλον μια λύση με την υπόθεση αυτή. Επίσης, η συγγήτρια μίλησε και για μια απόφαση του δικαστηρίου σε ό,τι αφορά τη δική μου πρόσληψη και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε ε, για τη χειρία μια θέση και τα λοιπά, για το διαγωνισμό που έγινε. Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Πρέπει να σας πω ότι με βάση προηγουμένων που υπήρχαν η ακύρωση μιας θέσης, ε, μια, χειρίας μιας θέσης, δεν σημαίνει και ακύρωση ορισμού. Ο κύριος Μπρούνο ήταν ένα καλό παράδειγμα, πρώην Γενικός Διευθυντής της Όλαφ. Ακυρώθηκε η ανακοίνωση της χειρίας της δικής του θέσης, παρέμεινε στη θέση του όμως. Η Επιτροπή, πρόεδρος Επιτροπής, έλαβε πάρα πολλές νομικές συμβουλέ και εξωτερικές από τρεις ξεχωριστούς εμπειρογνώμονες, τρεις διαφορετικές γνωμοδοτήσεις και την επίσημη επίση νομική γνωμοδότηση των υπηρεσιών Κοινοβουλίου Κομισιών και Συμβουλίου. ίδια ήταν η απόφαση ότι δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται με τον τρόπο αυτό η απόφαση αν υπάρχει ακύρωση του λεγόμενου vacancy notice. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση των, όλων των γλωσσών σε αυτές τις κοινοποιήσει. Και για να διευκρινιστεί εντελώ η κατάσταση, υπήρξε ανταλλαγή αλληλογραφίας με τους μόνιμους εκπροσώπους, ε, μόνιμους αντιπροσώπους Ιταλίας και Ισπανίας, με την πρόεδρο της ε, ΕΟΚΕ και μετά έληξε το θέμα. κάλεσα την κυρία Γιάλα να έρθει στην Επιτροπή μα. Το φάκελο μπορώ να τον διαθέσω ευχαρίστω πάντω για να δει από μόνη τη. Ήταν ενδιαφέρουσα η κατάσταση, το ομολογώ. Όσε πληροφορίε χρειάζεται η συγγήτρια, ευχαρίστω να τι τις διαβιβάσω. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα του κυρίου Βόν, τον ευχαριστώ για το ερώτημα αυτό γιατί μου θύμισε κάτι που ξέχασα. Να αναφέρω ένα άλλο αίτημα ε, στο ψήφισμα απαλλαγή του 2009 που αφορούσε τη δήλωση των οικονομικών συμφερόντων των μελών. Με τα χαράς μπορώ να σας ενημερώσω ότι η Επιτροπή μας πλέον τηρεί πλήρων, πλήρως τη σύσταση ε, που περιλάμβανε αυτό το ψήφισμα περί απαλλαγής. Να πω στον κύριο Βόν ότι ο αντιπρόεδρος που έχει τη σχετική αρμοδιότητα για τα δημοσιονομικά θέματα, ο κύριος Κράτσεκ, και εγώ συνεργαστήκαμε για να κάνουμε μια μεταρρύθμιση σε βάθος των δομών και διαδικασιών. Και νομίζω ότι έχουμε πλησιάσει όσο περισσότερο μπορούμε στην πλήρη διαφάνεια. Όχι ότι δεν είχε διαφάνεια και δεν υπήρχε υγεία, αν θέλετε, και ευρωεστία οικονομική στην Επιτροπή μας, απλά πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Και έρχομαι στο ερώτημα της κυρίας Ιβάνου για την αναφέρωση των δαπανών. Πράγματι υπήρξε ε, μια φυσική επανεξέταση και αναθεώρηση του προπολογισμού σε σχέση με το σχέδιο κατάσταση του προπολογισμού του 2012 με μια υποομάδα τη Επιτροπής Προπολογισμών η οποία εξέτασε εντελεχέστατα όλες τις δαπάνες. Το ίδιο εγχείρημα θα γίνει και σε σχέση με τον προπολογισμό του 2013. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό που πάντοτε προσπαθούμε να ε, πετύχουμε είναι εξοικονόμηση πόρων. Να σας δώσω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Ο Δόκτωρ Γκαλέα, το μέλο του συνεδρίου, ήρθε στην Επιτροπή μας πρόσφατα και από αυτόν και από τις υπηρεσίε του μάθαμε τις ε, οικονομίε που κατάφεραν να πετύχουν στο ελεκτικό συνέδριο με τις ε, ρυθμίσεις και τους διακανονισμού στον τομέα τη ασφάλειας. Με τον διευθυντή ε, τη υλικοτεχνική υποδομή, logistics, θα δώσει στο Λουξεμβούργο πώ μπορούμε και εμεί να πετύχουμε κάποια περαιτέρω εξοικονόμηση. Ο ομόλογό μου, ο κύριο Στάλ, πρέπει να πω ότι σίγουρα και αυτό θα πρέπει ε, να συμμετέχει, γιατί είναι στι κοινέ υπηρεσίε η ασφάλεια. Είναι ένα παράδειγμα όμω των προσπαθειών μα για εξοικονόμηση πόρων. Σε ό,τι αφορά ε, τα όσα είπε ο κύριο Σέπινγκ, η Επιτροπή μα για το 2012, αν λάβετε υπόψη τον πληθωρισμό, έχουμε αρνητική αύξηση αρκινητική ανάπτυξη μάλλον. Και μάλλον θα έχουμε και για το 2013 έναν προϋπολογισμό αρνητική ανάπτυξη. Πρέπει να σας πω, όπως το προείπα άλλωστε, ότι τον περισσότερο χρόνο τους ε, ε, τα μέλη μας ε, τον περνούν στις οργανώσεις τους και ξέρουν από πρώτο χέρι πώς βιώνει ο κόσμος την κρίση. Και γι' αυτό θα υποβάλουμε μια πολύ λογική πρόταση για τον προβλησμό του 2013 που θα απηχεί την πραγματικότητα το, το τι βιώνει ο κόσμος. Αναφέρεται επίσης στην αύξηση των προπλησμών επικοινωνίας των δύο επιτροπών. Αν έχει γίνει αυτό, αυξήσαμε δηλαδή τις επικοινωνικές μας δραστηριότητες, είναι γιατί το κάναμε γιατί να υπάρχει μεγαλύτερη προβολή, να είναι πιο γνωστές οι δραστηριότητές μας. Η συγγήτρια μίλησε και για την συμβολή μας στην νομοθετική διαδικασία και τη δημοσιονομική διαδικασία. Αναφέρατε και τον κύριο Ρεγκάλντο. Την προηγούμενη εβδομάδα το εφετείο του Βελγίου τον ε, απάλαξε από κάθε κατηγορία. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έχουμε. Εγώ ε, μπαίνω και στο facebook και γράφω σε blog. Τώρα με το Twitter δεν ασχολούμαι ενεργά, είμαι μάλλον παθητικός χρήστης ε, λόγω της δουλειάς που έχω ο αντιπρόεδρός μας για την επικοινωνία, η Άννα Μαρία Νταρμάνιν, είναι όλη την ώρα στο Twitter μπορώ να σας πω. Είναι από, τους πλέον, από τις πλέον ένθερμες ε, θειασότριες του είδους. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Μέλλον της Ευρώπης, ο Νικολάη Βάμιν, Δανός Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, είχε έρθει στην Ολομέλεια ε, την προηγούμενη Πέμπτη στην ΕΟΚΕ και μας μίλησε και μας είπε ότι εν καιρό οικονομικής και κοινωνική κρίση, κρίσης ο ρόλος τη επιτροπή σα είναι πιο σημαντικός από ποτέ, έτσι γιατί μιλήσατε εσεί για την ε, Δανή ε, Πρωθυπουργό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις θα περάσουμε ίσω στο Twitter να συνεχίσουμε. Λοιπόν, ο κύριος Χάρντεν από την Επιτροπή του Ευρωπαίου Διαπρέμιου Στολιτευτή έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. In uh, Ανταποκρινόμενο στην ερώτηση της κυρίας Γκρέσλερ όσον αφορά τον ακριβή αριθμό προσωπικού, έχουμε τις πληροφορίες. Είναι μια φωτογραφία που θα σας δώσουμε σήμερα θέτες καταστάσεω για το 2011 και θα στείλω τις πληροφορίες στην κυρία Γκρέσλερ μετά τη συνεδρίαση. η ερωτήση της κυρίας Αγιάλα Σέντερ, της εισηγήτριας, εστιάστηκε στο το θέμα του χρόνου. Πόσο χρόνο χρειαζόμαστε να εξεραστούμε τις διάφορες διαμαρτυρίες, καταγγελίες. Ας το δούμε αυτό από δύο πλευρές. Πρώτη πλευρά. Πρέπει να πετύχουμε ισορροπία. Μεταξύ του πόσο προσεκτικά ερευνούμε, σε τι βάθος μπαίνουμε και πόσος χρόνος χρειάζεται από την άλλη. Η ταχύτητα δεν είναι πάντα η βέλτιστη λύση. Καμιά φορά χρειάζεται χρόνος για να αντιμετωπιστεί μια υπόθεση. Στο αναγκαίο βάθο. Γνωρίζουμε όμως ότι όταν καθυστερεί δικαιοσύνη είναι σαν να μην αποδίδεται. Και πολλοί αναφερόμενοι θέλουν γρήγορη απόφαση. Και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε δεόντως θέλουμε να παρέχουμε διάφορες δυνατότητες για να χρησιμοποιούμε την ορθή διαδικασία για κάθε περίσταση και την ταχύτερη δυνατή. Η άλλη πτυχή. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις μπορούν να συμβούν και στο γραφείο του συνηγόρου του πολίτου, όπως και σε άλλες περιπτώσεις. Καθημερινά προσπαθούμε, επαγρυπνούμε, προσπαθούμε να αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, να ε, αναμένουν υποθέσεις που θα μπορούσαν να διεκπαιρεωθούν. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε ε, τις καθυστερήσεις άλλων ε, θεσμικών οργάνων όταν καθιστούν να μας απαντήσουν. Αλλά αυτά που συμβαίνουν εντός των υπηρεσιών μας προσπαθούμε να τα ελέγξουμε και να αποφύγουμε τις καθυστερήσεις. Στο ετήσιο σχέδιο μας έχουμε συμπεριλάβει βασικούς δείκτες που σχετίζονται με τον χρόνο ε, επεξεργασίας υποθέσεων. Ένα δίκτυ θα ήθελα να αναφέρω. Αυτός αφορά το χρόνο που χρειάζεται για το να κριθεί αποδεκτή μια υπόθεση. Θα ξεκινήσει έρευνα ο διαμεσολαβητής για αυτή την υπόθεση ή είναι εκτός των δικαιοδοσιών του ή για κάποιον άλλο λόγο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η υπόθεση. Έχουμε θέσει στόχο στο ετήσιο διαχειριστικό μας σχέδιο Θέλουμε η απόφαση να λαμβάνεται εντό μηνό. Και αυτό να γίνεται στο 90% των υποθέσεων. Πέρσι δεν τα καταφέραμε. Καταφέραμε 70%. Εξετάσαμε τι βελτιώσει θα μπορούσαμε να επιφέρουμε. Τον ίδιο στόχο έχουμε θέσει και το 2012, το 90%. Προσπαθήσαμε να βρούμε τρόπους για να βελτιωθούμε και ένα κομμάτι της εσωτερικής αναδιοργανώσεως που προανέφερα έχει στόχο την επιβράχυνση, την βράχυνση μάλλον της διαδικασίας. Και αντί να απαντά προσωπικά δημοσιολαβητή να λέει στον αναφέροντα ότι δεν μπορώ να δεχτώ μια υπόθεση και σου δίνω την τάδε συμβουλή, ποιο σα μπορεί να σε βοηθήσει, αντί να γίνεται αυτό, θα λαμβάνω επιστολή που θα υπογράφει ο επικεφαλής του αρχείου μας, θα περνάει η διαδικασία ε, η διαδικασία θα είναι πολύ πιο σύντομη, οπότε οι πληροφορίες και οι συμβουλές θα χορηγούνται πολύ πιο γρήγορα στον αναφερόμενο. Ε, ελπίζω του χρόνου να μπορέσω να σας πω ότι έχουμε βελτιώσει σημαντικά το στόχο του 70%, τον έχουμε ξεπεράσει και πιστεύω ότι πράγματι ο στόχος του 90% είναι ρεαλιστικός. Για το 2012 έχουμε σχεδιάσει και αναβάθμιση των συστημάτων πληροφορικής. Έχουμε εξωτερικό σύμβουλο που την επόμενη εβδομάδα θα έρθει και θα εξετάσει τα συστήματα, τους υπολογιστές μας, θα κάνει συστάσεις για τη βελτίωση ε, του συστήματος του ολοκληρωμένου που έχουμε, της πληροφορικής. Τέλος, για να απαντήσω στα όσα αναφέρθηκαν για το Twitter. Πράγματι, αν δεν υπάρχει στα κοινωνικά μέσα, δεν υπάρχει. Ένα κομμάτι του ρόλου του διαμεσολαβητή είναι η επικοινωνία με τους Ευρωπαίους πολίτες με τον αποτελεσματικότερο τρόπο και ένα άλλο σχέδιο που έχουμε για το 2012 είναι να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την ορατότητά μας στα κοινωνικά μέσα συμπεριλαμβανομένου και του Twitter. Το 2012 λοιπόν πρέπει να είναι ο χρόνος κατά τον οποίο θα μπει στο Twitter ο διαμεσολαβητής και θα τουιτάρει. Ευχαριστώ κύριε Χάρντεν. Και τέλος, εξίσου σημαντικός φορέας, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εποπτική Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων. Ερώτηση. Είναι ασφαλή τα στοιχεία μας στο Facebook και σε άλλα κοινωνικά μέσα. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε εδώ. Ίσως μπορείτε να απαντήσετε εν συντομία όμως, διότι έχουμε καθυστερήσει. Ίσως λοιπόν μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Εξετάζουμε τη στρατηγική επικοινωνία μας και ίσως και εμείς φέτος ξεκινήσουμε να τουιτάρουμε. Αλλά υπάρχει πρόβλημα με το Facebook όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, οπότε δεν είμαστε σίγουροι ότι θα το χρησιμοποιήσουμε το Facebook. Πολλές ερωτήσεις ετέθησαν σε τέσσερις κατηγορίες. Πρώτα απ' όλα δήλωση αξιοπιστίας 2009-2010. Υπάρχει ένας υπεύθυνο για επικοινωνία για το λογιστικά και υπάρχει ένας υπεύθυνο για τον εκ, ε, έλεγχο. Δεν ξέρω ποια είναι η γαλλική έκφραση. Τέλος πάντων, κάποιος είναι ανεξάρτητος από το τμήμα τη Διεύθυνση Οικονομικών, ανεξάρτητος σύμβουλος που εργάζεται σαν επιθεωρητής ε, ε, ελέγχου δεδομένων, προστασία δεδομένων, που εκτελεί αυτό το καθήκον του 2011. Δημιουργήσαμε το Μητρό Εξαιρέσεων που είναι διαθέσιμο και για τη χρήση 2010 και 2011. Και τέλος, όσον αφορά τα οικογενειακά επιδόματα, έχουμε συστήσει να δημιουργήσει ένα σύστημα. Παρακολουθούνται και ελέγχονται μία φορά το χρόνο αυτά ε, μέσω ειδικού εντύπου που έχουμε θεσπίσει για αυτό το σκοπό. Για τα KPIs, τρίτο ερώτημα. Στο δεύτερο ήμιση του έτους θα το αναπτύξουμε αυτό μετά τα αποτελέσματα των εξωτερικών διαβουλεύσεων. Θέλουμε να αναπτύξουμε πρώτα στρατηγική και προτεραιότητες όσον αφορά τους δείκτες επιδόσεων Θέλουμε τους βασικούς δείκτες επιδόσεων ή KPIs να αναπτύξουμε για να κάνουμε τις δέουσες μετρήσεις. Ε, τι συνέχεια δίνουμε στις συστάσεις. Θέλουμε οι συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εντάσσονται σε ειδικό κεφάλαιο το ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του 2011. Ετέθη ένα ερώτημα για τα ηλεκτρονικά συστήματά μας. Το έχει θέσει και ο δικός μας εσωτερικός έλεγχος. Συμφωνούμε απόλυτα. Χρειάζεται και το χρειαζόμασταν από καιρού αυτό ένα αποτελεσματικό σύστημα για την επεξεργασία και προστασία των ευαισθητών δεδομένων. Σημειώστε ότι το EDPS βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, ο φορέας μας βασίζεται για την υποδομή μα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι αντιμετωπίσαμε. Υπήρχε αμφιβολία κατά πόσο μπα χρησιμοποιήσουμε τι συμφωνίε πλαίσιο για την πληροφορική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τόσο μεγάλο πρόγραμμα. Υπογράψαμε τώρα λοιπόν. Ανανεωθεί συμφωνία διοργανική για συνεργασία με το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για άλλε πτυχέ. Και στο πρωτόκολλο αναφέρεται σαφώ ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, συμφωνίε πλαίσιο για την πληροφορική διότι διαφορετικά είμαστε πολύ μικροί για να διοργανώσουμε κάτι τέτοιο για να προτεστούμε. Το 2011 κάναμε εξολόγηση της αγοράς, επιλέξαμε ανάδοχο, λογισμικό, όλα έχουν υπογραφεί, ξεκινήσαμε και το σύστημά μας θα δοκιμαστεί και θα είναι έτοιμο μέχρι το Μάιο φέτος. Πριν εισάγουμε τις πληροφορίες μας, θα κάνουμε εσωτερικό έλεγχο και εξωτερικό έλεγχο επί του αναδόχου για να είμαστε βέβαιοι ότι το σύστημα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσει που έχουμε όσον αφορά την ασφάλεια. Τέλος, ο διαγωνισμός. Οι διαγωνισμοί αναφερθήκαν το λεκτικό συνέδριο. Ήταν παρατήρηση και ουχή σύσταση. Σας αποστήλαμε κύριε Πρόεδρε και στην εισηγήτρια πλήρη απάντηση στην παρατήρηση. παρόδο ότι αποδεχόμεθα πλήρω την παρατήρηση του ελεγκτικού συνεδρίου. Δηλαδή, ότι οι εσωτερικοί διαγωνισμοί δεν είναι συνηθισμένη πρακτική. Η καλύτερη πρακτική είναι η χρήση της υπηρεσίας ΕΨΟ. Οι διαγωνισμοί που έλαβαν χώρα χρησιμοποίησαν και οι δύο την ΕΨΟ και στην πλήρη απάντηση θα δείτε γιατί στι εξαιρετικέ περιστάσεις που επεκράτησαν το 2009 που αφορούσε ότι θα χάναμε το μισό προσωπικό μας που ήταν με ε, συμβάσεις ορισμένης διαρκείας, ε, έπρεπε να το κάνουμε αυτό για να έχουμε εσωτερική ε, ισορροπία. Ήταν εξαιρετική περίσταση και γι' αυτό οργανώσαμε εσωτερικούς διαγωνισμούς, αλλά έχετε την πλήρη απάντηση. Ευχαριστώ τον κύριο Τόξη και όλους τους εκπροσώπους των άλλων θεσμικών οργάνων. Ολοκληρώνεται εδώ αυτή η συζήτηση και μπορώ να δώσω το λόγο στον κύριο Λουγκαλία, τον εκπρόσωπο του Ελεκτρικού Συνεδρίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, όπως και προλαλήσαντες, να σας συγχαρώ θερμά για την εκλογή σας στη θέση του Πρόεδρου της Επιτροπής έλεγχο του προπολογισμού. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Είμαι βέβαιος ότι και ο πρόεδρος και οι συναδελφοί μου από το Ελληνικό Συνέδριο προσβλέπουν να σας, να σας γνωρίσουν καλύτερα, να συνεργαστούν μαζί σας και με τα μέλη της Επιτροπής σας, ώστε να έχουμε την καλύτερη ε, και τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία των εργασιών σας εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω και την ε, εισηγήτριά σας, την κυρία Γιάλα Σέντερ, την οποία πρέπει να πω ότι θαυμάζω για την αφοσίωση, τη δέσμευσή της. Παρακολουθεί το έργο του ελεγκτικού συνεδρίου για να υπάρξει μεγαλύτερη λογοδοσία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Να ευχαριστήσω επίσης και όλους τους βουλευτές που υπέβαλαν ερωτήματα και έγγραφα αλλά και προφορικά σήμερα σε σχέση με τη διαδικασία απαλλαγής. Επιτρέψατε μου κύριε Πρόεδρε να τονίσω την ε, συνεργασία που πράγματι είχαμε με όλους τους γενικούς γραμματείς ε, των οργανισμών που συζητήσαμε σήμερα το πρωί. Νομίζω ότι είναι σε βελτίωση. Ε, υπάρχει μεγαλύτερη, πιο χρηστή οικονομική διαχείριση και πολύ καλύτερος έλεγχος και παρακολούθηση των συστάσεων και παρατηρήσεων που διατυπώνουμε εμείς στις εκθέσεις μας. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σημειώσαμε τα σημαντικά στοιχεία και επιχειρήματα των εκπροσώπων των διαφόρων οργανισμών και τις απαντήσεις που έδωσαν σε ερωτήσεις. Πρέπει να σας πω ότι θα συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε, να ελέγχουμε, να παρακολουθούμε τα διάφορα γυρώμενα ζητήματα και οτιδήποτε άλλο προκύψει και σχετίζεται με τη χρηστή οικονομική διαχείριση στον διοικητικό ε, τομέα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much, uh, Mr. I think... Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκαλέα. Εδώ νομίζω είναι το σωστό σημείο να σας ευχαριστήσω και εσάς και το ηλεκτρικό συνέδριο που σεβόμενοι την εξαρτησία και των δύο θεσμικών οργάνων χρειαζόμαστε πάντα τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού συνεδρίου. Θέλω τώρα να δώσω το λόγο πάλι στην εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να πω απλά ότι είμαι πολύ ικανοποιημένη. Ίσως κάποια θέματα που δεν απαντήθηκαν διμερώς ε, στη συνεργασία που έχουμε θεσμικών θα μπορούσαν να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γκαλέ για την δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα και τον, να του εκφράσω και εγώ το θαυμασμό μου. Είναι αμοιβαίο. και όλους τους εκπροσώπους ε, που ήταν εδώ θέλω να τους ε, ευχαριστήσω προσωπικά τον καθένα. Ελπίζω να έχουμε και κάποια γυναίκα γενική γραμματέα σύντομα στην παρέα. Ολοκληρώνοντας, αν μου επιτρέπετε, να ευχαριστήσω όλος ιδιαίτερο τη γραμματεία της Επιτροπής μας. Μπορεί να την γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ακόμα, αλλά θα τη μάθετε. Και θα δείτε ότι χωρίς την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε τη γραμματεία δεν θα μπορούσαμε να εργαστούμε. Να ευχαριστήσω και την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου που με διαφώτισε σε πολλές περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση του σημείου αυτού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας από τα άλλα θεσμικά όργανα. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο, σημείο 9 της ημερησίας διάταξης. Ειδική έκθεση Είναι σωστό ο συνδυασμό στη διαχείριση των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων. Η συγγήτρια η κυρία Σουζάνα Προσμποχατά. Και από το Ελληνικό Συνέδριο χαιρετίζω τον κύριο Ολάβη Αλα Και θα ήθελα να του δώσω αμέσως και το λόγο. Κύριε Ολάβη Αλανίσιλε, έχετε το λόγο. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω ίσως οι συζητήσεις που γίνουν αυτή τη στιγμή ε, μέσα στην αίθουσα να μετατοπιστούν εκτός της αίθουσας για να μπορέσουμε να συζητήσουμε με την ημερησία διάταξη. Κυρία Άλλα Νησιλέ, έχετε το λόγο. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές κυρίες και κύριοι. Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζω σήμερα την ειδική έκθεση του συνεδρίου για την γεωργοπεριβαλλοντική στήριξη. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας δώσω κάποιες πληροφορίες σε σχέση με την γεωργοπεριβαλλοντική στήριξη και να εξηγήσω το πεδίο εφαρμογή του ελέγχου μας. Κατά δεύτερον θα σας παρουσιάσω τα κύρια πορίσματα του συνεδρίου και τα βασικά του μηνύματα και αν κατακλείδη θα επισημάνω ορισμένες από τις βασικές μας συστάσεις η γεωργοπεριβαλλοντική στήριξη είναι πάρα πολύ σημαντική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ του κοινοτικού προπολογισμού δαπανώνται για την πολιτική αυτή ετησίω. Και πρόκειται για αντιστάθμιση σε περίπου, μάλλον σε αποσμίωση σε περίπου 600.000 αγρότε ε, για το επιπρόσθετο κόστο ε, και, και τα έσοδα τα οποία ενδεχομένω χάνουν σε σχέση ε, με τις περιβαλλοντικά φιλικές γεωργικές πρακτικές πρέπει να εφαρμοστεί η πολιτική αυτή με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι μια πρόκληση. Η Γιώργο περιβαλλοντική πολιτική είναι θελοντική για τους ε, αγρότες. Επομένως θα πρέπει να είναι ελκυστικό το επίπεδο των πληρωμών σε σχέση με τις δεσμεύσεις που πρέπει να αναλάβουν και το κόστος που θα πρέπει να επομιστούν οι αγρότες. Και από την άλλη πλευρά οι πληρωμές θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στο επιπλέον κόστος συν το πιθανό κόστος συναλλαγών, συναλλαγής, transaction costs. Θα πρέπει λοιπόν για να συμμετέχουν οι αγρότες στην πολιτική αυτή να μην έχουν χρηματοοικονομικό όφελος. Σε σχέση με το πεδίο εφαρμογή. θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι στόχος του ελέγχου ήταν να δει κατά πόσον ε, ε, η γεωργοπεριβαλλοντική στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καλά σχεδιασμένη και έχει τη σωστή διαχείριση. Ένα από τα ερωτήματα ε, στη διάρκεια του έλεγχου αυτού που κληθήκαμε να απαντήσουμε είναι κατά πόσο είναι σχεδιασμένη η πολιτική αυτή για να δίνει απτά περιβαλλοντικά ε, αποτελέσματα. Δεν προσπαθήσαμε όμως με τον έλεγχο αυτό καθεαυτό να μετρήσουμε, να ποσοτικοποιήσουμε τον αντίκτυπο της ε, στήριξης αυτής ε, για το περιβάλλον. Δεν σας ε, παρουσιάσω τα πορίσματα, τα βασικά πορίσματα, να σας πω σαν γενική παρατήρηση ότι υπήρξε σημαντική πρόοδος στη διάρκεια αυτών των 20 ετών από την εισαγωγή της πολιτικής αυτής. Πολλοί αγρότες πλέον υλοποιούν, εφαρμόζουν πιο βιώσιμες πρακτικές δεν θα το έκαναν χωρίς αυτή την υποστήριξη. Πάντως, ε, διαπιστώσαμε σε τομείς διάφορους ότι πρέπει να γίνουν ε, βελτιώσεις. Τρία πορίσματα θέλω να σας επισημάνω. Πρώτον, γενικά οι στόχοι ήταν ασθενείς, αδύναμοι, ε, μάλλον ε, συγγνώμη, ας, ασαφείς, αόριστοι και δεν ήταν δυνατόν επομένως να αξιολογήσουμε το βαθμό στον οποίο επετέχθησαν αυτοί οι στόχοι. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι η πολιτική δεν έχει σχεδιαστεί, ούτε έχει παρακολουθηθεί ως προς το κατά πόσο να αποδίδει απτό περιβαλλοντικό όφελος. Δεύτερον, υπήρξαν προβλήματα, σημαντικά προβλήματα, παρότι υπήρξε καλή ε, καθοδήγηση προς τους ε, αγρότες, υπήρξαν πάντως σημαντικά προβλήματα σε ό,τι αφορά τα ποσά ε, των ενισχύσεων. Υπήρχαν αδυναμίες και προβλήματα με τους υπολογισμούς και δεν υπήρχε διαφοροποίηση ανάλογα με τις συνθήκες που επικράτουν σε περιφερειακή τοπικό επίπεδο. Κατά τρίτον, τα κράτη-μέλη πρέπει να διαθέτουν την υποστήριξη αυτή σε σχέση με τις ειδικές ανάγκες. Ο έλεγχος που κάναμε όμως κατέληξε στο ότι τα κράτη-μέλη δεν είχαν επαρκώς λάβει υπόψη τους ε, τον ε, επαρκή βαθμό στόχευσης στις συγκεκριμένες ανάγκες. Δεν είχαν κάνει δηλαδή κόστου ε, κόστους-οφέλους. Με βάση τον έλεγχό μας προβήκαμε σε μια σειρά από για τη βελτίωση της υλοποίησης της γεωργοπεριβαλλοντικής υποστήριξη, Θα σα αναφέρω μερικέ από αυτέ. Η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι στα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου θα εφαρμόζονται και θα τίθενται σαφείς στόχοι και θα είναι αιτιολογημένη διασύνδεση μεταξύ περιβαλλοντικών πιέσεων και γεωργοπεριβαλλοντικών πληρωμών. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συλλέγουν και να αναφέρουν αξιόπιστα σχετικά επίση με το αντικείμενο δεδομένα σε ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό όφελο και να τα χρησιμοποιούν στου σκοπού τη παρακολούθηση. Για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού κομισιών θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει πιο εστιασμένη στόχευση των δαπανών στι ειδικέ περιβαλλοντικέ ανάγκε. Σημειώσαμε ότι η νέα γεωργική νομοθεσία που προτείνει η Κομισιόν προσπαθεί να αντιμετωπίσει εν μέρη τις συστάσεις μας. Δηλαδή, ε, για παράδειγμα, προτίθεται να δημιουργήσει ένα νέο ξεχωριστό μέτρο για την βιολογική, την οργανική γεωργία, για να υπάρχει μεγαλύτερη ορατότητα. Σε σχέση λοιπόν με τη σύσταση παριθμών 4 που έχουμε διατυπώσει, δηλαδή ότι η Κομισιόν θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον οι γεωργοπεριβαλλοντικέ πληρωμέ θα πρέπει να υποδιαιρεθούν σε απλέ, γενικευμένε γεωργοπεριβαλλοντικέ δράσει και πιο απαιτητικέ, more demanding δράσεις και είχαμε πει ότι η στήριξη της ε, βιολογικής γεωργίας θα πρέπει να συνιστά ένα ξεχωριστό μέτρο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι συλλογικέ συμβάσει, όπου μα έλαβε υπόψη η Κομισιόν. Θεωρούμε ότι η προσέγγιση σε ορισμένε υποθέσει, περιπτώσει είναι πολύ σημαντική αυτή η προσέγγιση, αν θέλουμε να πετύχουμε του περιβαλλοντικού στόχου. Η καλύτερη στόχευση πάντως από τα βασικά θέματα παραμένει μια σημαντική πρόκληση για την ε, λήψη αποφάσεων και για την υλοποίηση νέων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξη. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ για την προσοχή σας. Να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια, την κυρία Μπρος Μποχάτα, για το έργο της και τα επικοδομητικά της σχόλια και συστάσεις. Με τα χαρά θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Αλανίσελε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία εισηγήτρια τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω καταρχήν τη δική μου γνωμοδότηση για την ειδική αυτή έκθεση ε, Όσον αφορά την ε, ε, αποτελεσματικότητα των γεωργικών περιβαλλοντικών ενισχύσεων, θα ήθελα επί ευκαιρία να εξετάσουμε τα αποτελέσματα. Γιατί η γεωργοπεριβαλλοντική ενίσχυση είναι ένα σημαντικό τμήμα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν 22 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται ε, για την ενίσχυση αυτή και σαν τμήμα της ανάπτυξης της υπαίθρου. Η Κομισιόν εγκρίνει τα προγράμματα που, εγκρι... προετοιμάζουν τα κράτη-μέλη και ο στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι να δοθούν κίνητρα στους ε, παραγωγούς, χειρουργούς παραγωγούς, να χρησιμοποιούν περιβαλλοντολογικά βιώσιμες λύσεις. Ε, μετά η Κομισιόν συνάπτει συμβάσεις με τα εν λόγω κράτη-μέλη που αναλάβουν την υποχρέωση να, αναλάβουν, να εφαρμόσουν συγγνώμη, τις ε, προβλεπόμενες πρακτικές. Κατόπιν η Κομισιόν ελέγχει αν τα αποτελέσματα για το περιβάλλον ήταν πραγματικά απτά και θετικά. Από τότε που εισηχθεί αυτή η μέθοδος ε, επιτέχθη σημαντική πρόοδος, παραμένουν όμως σημαντικά προβλήματα που μειώνουν την επίδραση των ολογομέτρων. Θα σας πω ποιες είναι αυτές οι ελλείψεις. Σύμφωνα με το Ελεκτικό Συνέδριο, η πολιτική αυτή δεν έχει εφαρμοστεί και ελεχθεί κατά τέτοιο τρόπο τους ώστε τα αποτελέσματα είναι πραγματικά απτά, γιατί δεν είναι δυνατόν να τα μετρηθούν αυτά τα αποτελέσματα και αυτό δεν μπορούν να ελεγχθούν σωστά. Επίσης θα πρέπει η αιτιολόγησή τους να είναι καλύτερη. Είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί δηλαδή η εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Και γι' αυτό και εδώ συμφωνώ με το ηλεκτρικό συνέδριο, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν καλύτερα οργανωμένα, καλύτερα εστιασμένα προγράμματα που να ελέγχονται περισσότερο πριν από την εγκρισή τους. Αυτή η πολιτική θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις ειδικέ ανάγκες για την περιβαλλοντολογική προστασία. Είναι απαράδεκτο το 39% των περιπτώσεων που στοιχεία πρασινίσματος του ΣΥΠΗΝ που εμπεριέχονται. Ε, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη ευελιξία. Ε, υπάρχει ένα μενού επιλογής ε, δυνατοτήτων και λύσεων που προβλέπεται και προτείνεται και το θέμα είναι κατά πόσο θα πρέπει να επιβάλλονται τα μέτρα εκ των άνω προς τα κάτω. Βέβαια, ίσως κάποιες επικρίσεις που ακούστηκαν στο Συμβούλιο να είναι βάσιμες. Τα κράτη-μέλη ε, πώς θα κινηθούν όμως. Ευχαριστώ την εισηγήτρια που τα αναφέρει το σημείο αυτό στην έκθεσή της. Λοιπόν, ακούγονται διάφορες απόψεις και εκφράζονται και τοποθετήσεις ε, από πλευράς του ελεκτικού συνεδρίου σχετικά με τις αγροπεριβαλλοντικές πτυχές. Ε, χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν σωστά τα 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας. που διατίθενται λοιπόν στον τομέα αυτό. Και πιστεύω ότι ένα από τα προβλήματα που θα πρέπει να επιληθούν και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό. Τα συμπεράσματα της 13ης Δεκεμβρίου του Συμβουλίου ε, πρέπει να ληφθούν υπόψη. Συζητήθηκε η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξε κάποια συμπεράσματα Λοιπόν, ε, υπογραμμίζεται τελικά ότι πρέπει να έχουν συγκεκριμένο στόχο. Η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου αναφέρεται σε σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί και τα πραγματικά αποτελέσματα θα είναι μακροπρόθεσμα ορατά. Με άλλα λόγια, το Συμβούλιο το Συμβούλιο είναι τυφλό, δεν καταλαβαίνει ποια είναι τα συμπεράσματα στο οποίο καταλήγει το ηλεκτρικό συνέδριο και θεωρώ Νομίζω ότι δεν έχουμε κανένα εκπρόσωπο της, ε, του Συμβουλίου εδώ, κακός, αλλά θα ήθελα να μου ακούσω το Συμβούλιο να μας πει πώς καταλήγει σε αυτά τα συμπεράσματα μετά από τόσο επικριτική μελέτη του ηλεκτρικού συνεδρίου και αν δεν είναι παρόν το Συμβούλιο, ίσως θα μπορέσουν να μας δώσει την απάντηση αυτή γραπτά. Πώς μπορεί να υπάρχει τεράστια αυτή η διαφορά μεταξύ της έκθεσης του ηλεκτρικού συνεδρίου και των συμπερασμάτων στα οποία καταλήγει εξ αυτών το Συμβούλιο. Λοιπόν, Πρόεδρε, μπορώ απόλυτα να συμφωνήσω με τα συμπεράσματα της εισηγήτριας. Με ενδιαφέρεται πολύ η φύση και το περιβάλλον, αλλά έχω την εντύπωση, εάν τα προβλήματα αυτά εφαρμόζονται κατά τέτοιο τρόπο, θα πρέπει να τα εξετάσουμε πάρα πολύ ε, επικριτικά και να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Διαφαίνονται βέβαια κάποια θετικά παραδείγματα, θετικά σημεία που βλέπουμε πώς ε, πραγματικά οι παραγωγοί αποτελεσματικά χρησιμοποιούν τα χρήματα αυτά αλλά θα πρέπει να δούμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούν να παίρνουν μόνο τα χρήματα, θα πρέπει να τηρούν και τα κριτήρια στα οποία βασίζεται η χορήγηση των χρημάτων αυτών. Αν δεν το κάνουν, δεν θα μπορούμε να προχωρήσουμε σωστά έτσι. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Δεν έχει κανένα άλλο συζήτηση το λόγο, εκτό αν παρέβλεψα κάποιον. Όχι. Οπότε θα μπορούσα να ξαναδώσω το λόγο στο ηλεκτρικό συνέδριο. Äh, Α, συγγνώμη, η Κομισιόν που ήθελε να τοποθετηθεί από αυτόν. Bitte. <laughs> Yeah, you're welcome. The floor Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεκτικό συνέδριο και την εισηγήτρια για τα σχόλιά τους και για τις συστάσεις τους. Τονίζεται η πρόοδος επιτεύχθη. Ευχαριστούμε το ελεκτικό συνέδριο για τις συστάσεις που έκανε. Πρόεδρε, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία που έχουν οι περιβαλλοντικές πτυχές για την ΚΑΠ. Αναγνωρίζουμε τη σημασία που έχει διότι το 25% των ενισχύσεων των αγροτικών που χρησιμοποιούνται αφορούν τα μέτρα που συζητούμε. Και όπως προανέφεραν τα μέλη, 25% του συνολικού προϋπολογισμού αφορά τα μέτρα αυτά. Έχει καταγραφεί πρόοδος. Όσον αφορά τις επικρίσεις, κάποια σχόλια έχω. Να απαντήσω σαφώς το τεθέν ερώτημα Την επόμενη περίοδο λοιπόν, 2014-2020, η ΚΑΠ θα ενισχύσει την πράσινη διάσταση. Καλύπτοντας και τους δύο πυλώνες. Στον πρώτο πυλώνα θα είναι γενικότερη εδαφική προσέγγιση. Ακολουθώντας τις διαπιστώσεις του ελεκτικού συνεδρίου και θα ληφθούν μέτρα που εφαρμόζονται ετησίως και εκπροσωπούν το 30% των κονδυλίων των αμέσων πληρωμών. Στο δεύτερο πυλώνα θα υπάρχουν πιο στοχευμένες προσεγγίσεις και θα πληρώσουμε αυτά που είναι πέρα από, το, από την βάση που έχει καθοριστεί από τα μέτρα του πρώτου πυλώνα. Αυτή η βάση θα ποικίλει κατά περίπτωση. Η βάση για την Ατούρα 2000, η βάση για την οδηγία για τα ύδατα, η βάση για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Θα διαφοροποιούνται όλα αυτά σε διαφορετικά επίπεδα απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον συνδυασμό των υποχρεωτικών απαιτήσεων για την ορθή γεωργική περιβαλλοντική προσέγγιση και τις συνθήκες που πρέπει να επικρατούν. Η βάση μεταβλητή λοιπόν θα λαμβάνει υπόψη τις επικρατούσες καταστάσεις και αυτό που θα εξακολουθούμε να πληρώνουμε θα είναι συμπληρωματικές δαπάνες κόστος συναλλαγής ε, πέρα από τις απαιτήσει της βάσης. Αυτή είναι η κατέθεση που θα ακολουθήσουμε. Ενίσχυση εστίασης στο δεύτερο πυλώνα και επιβάλλοντας τη νέα διάσταση του πρασινίσματος στον πρώτο πυλώνα. Όλα αυτά μαζί θα εφαρμοστούν και θα υπάρχει και έλεγχος. Πώς? Ενισχύοντας την αξιολόγηση και την εποπτεία. Θα τεθεί νέο πλαίσιο διάδοχο του υφισταμένου. Θα είναι κοινό έλεγχος αξιολόγηση, κοινό πλαίσιο. Κάτι που ήδη υπάρχει, που εφαρμόζεται από τον 60-98 τον κανονισμό για την ισχύουσα περίοδο και αυτός θα ενισχυθεί για να συμπεριλαμβάνει δείκτες που αφορούν τους δύο πυλώνες. Το κοινοτικό πλαίσιο, το κοινό πλαίσιο ελέγχου και αξιολογήσεως που υπάρχει, το SMIF, απαρτίζεται από δείκτες αποτελεσμάτων ροής και εκροής. Αυτό το πλαίσιο βεβαίως συμπεριλαμβάνει 7 δείκτες ε, συνεπειών, οι 4 καλύπτουν την περιβαλλοντική διάσταση. Νερό, έδαφος, βεπικιλότητα και τα λοιπά. Να το υπογραμμίσω ήθελα αυτό, διότι όταν προσμετρούμε τα αποτελέσματα της αγροπεριβαλλοντικής πολιτικής πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τον χρόνο για την προσμέτρηση των αποτελεσμάτων και των συνεπειών. Χρειάζεται χρόνος για να γίνει αυτή η αποτίμηση. Με τα χαράς Άκουσα το ελεκτικό συνέδριο να λέει ότι 16 χρόνια εφαρμογής της πολιτικής που ξεκίνησε από τον κανονισμό 2078 92, από το 92 μέχρι τώρα, απεκόμισε ωφέλη. Χρειάστηκε χρόνος. Ακολουθούμε σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται ενίσχυση αυτή η προσέγγιση. Το ξέρουμε. Συμφωνούμε με την εισηγήτρια και το ελεκτικό συνέδριο. Χρειάζονται βελτιώσει όσον αφορά τον έλεγχο της αξιολόγησης. Χρειάζονται καλύτεροι δείκτες στοχευμένοι, όχι μόνο στοχευμένα μέτρα, αλλά και στοχευμένοι δείκτες για αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολιτικής. Γι' αυτό έγιναν προτάσεις. Στις νέες προτάσεις ενισχύουμε το ρόλο του δικτύου για την αξιολόγηση, του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την αξιολόγηση που θα ενισχυθεί και οι προσπάθειες του δικτύου θα σχετίζονται με τις προσπάθειες άλλου δικτύου. Το δίκτυο για την ανάπτυξη της υπαίθρου και της σχετικής πολιτικής για να διαδώσουμε τις σωστές πληροφορίες προς τους γεωργούς και τις καλύτερες πρακτικές που υπάρχουν και συλλέγονται και διαβιβάζονται στο δεύτερο δίκτυο. Νομίζω ότι σωστό δρόμο ακολουθούμε και στη δεύτερη φάση θα κάνουμε ακόμα καλύτερες προσπάθειες. Τώρα, τις επικρίσεις που ακούστηκαν, θα ήθελα να τις αναφέρω, να αναφέρω κάποια στοιχεία. Οι περιβαλλοντικές πιέσεις που εντοπίστηκαν στην ανάπτυξη της υπαίθρωσης ειδικά προγράμματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μαζί με άλλα μέσα της ΚΑΠ που ήδη εφαρμόστηκαν Αναφέρομαι στο άρθρο 68 του κανονισμού για τις άμεσες πληρωμές. Και το στοιχείο της πολύμορφης συμμόρφωσης, της πολλαπλής συμμόρφωσης που θα υπογραμμίσω, και μέτρα που αναλαμβάνονται όσον αφορά τα απορροκυπευτικά και τα σχετικά προγράμματα εντός του πρώτου πυλώνα ε, την τρέχουσα περίοδο. Τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα ανταποκρίνονται και σε πιέσεις αλλά και σε δυνατότητες. Όπως τη δυνατότητα προστασίας ε, των υδάτων στις περιοχές συλλογή υδάτων, ε, διεύρυνση της βιοπικιλότητας, αύξηση της και επίτευξη βασικών στόχων που επιτυχάνονται μέσω των διαφόρων προγραμμάτων που εφαρμόζονται επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Λοιπόν, πρέπει να λάβετε υπόψη στι επικρίσει όταν ενέκρινε τα προγράμματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έλαβε υπόψη του ευφύ στόχου που παρουσιάζονται στα προγράμματα. Οι στόχοι είναι ευφύς, αλλά δεν είναι απλό στόχοι, αλλά συσχετίζονται και όταν μετρούμε προσπάθεια μιας πολιτικής, πρέπει να έχουμε υπόψη και τι συνδέσεις υπάρχουν μεταξύ στόχων προγραμμάτων που οδηγούν σε συνολική προσπάθεια για την επίτευξη αποτελέσματος. Τώρα λοιπόν, ήδη ανέφερα τον ελεγχό, θα ήθελα να αναφερθώ στην ανάγκη, μάλλον την επίκριση για τα ελάχιστα επίπεδα συμμετοχής που απαιτούνται ούσω ώστε να επιτευχθούν τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά αποτελέσματα. Τονίζεται το εξή στοιχείο. Κάνουμε υπολογισμό πρημοδοτήσεων. Βάσει συμπληρωματικών δαπανών και άλλων στοιχείων. Τον υπολογισμό τον κάνουμε μέσω των δύο παραμέτρων, δασικών παραμέτρων. Δεν βασιζόμαστε επί ποσού Βασιζόμαστε επί αντικειμενικών στόχων ε, στους υπολογισμούς. Είναι ευθύνη των κρατών μελών υπολογισμός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τον υπολογισμό κατά την έγκριση των προγραμμάτων. Λεπτομερέστατος είναι αυτός ο υπολογισμός. Απαιτεί τεχνογνωσία. Χρειάζονται πολλοί ανθρώπινοι πόροι. Εφαρμόζεται η κοινή διαχείριση συνεπώς. Και επομίζεται τις ευθύνες στο κράτος μέλος των υπολογισμών. Εξετάζει τον υπολογισμό Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητάει και συμπροματικέ πληροφορίε για αυτό το σκοπό από τα κράτη-μέλη. Πρόεδρε, το 39% που αναφέρεται των συμβάσεων που δεν συνδεόταν με συγκεκριμένες περιβαλλοντικές πιέσεις είναι κάτι που θέλω να υπογραμμίσω. Όχι, δεν λαμβάνονται υπόψη μόνο οι περιβαλλοντικές πιέσεις, αλλά αναλύοντας δυνατότητες όπως είναι η βιοπικιλότητα ή τα, η χώρη συλλογή υδάτων και αυτές οι πτυχές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Οι λεκάνες απορροής. Άρα, αν δεν ακολουθεί το αυτή η προσέγγιση μέχρι τώρα, ίσως θα είχαμε μεγαλύτερη κατάληψη γεών Όσον αφορά τη συλλογική προσέγγιση, ναι, υπάρχουν νέες προτάσεις για να ενισχυθεί η διάσταση της συλλογικής προσέγγισης. Συνεργασία χρειάζεται. Και ποιος θα ηγείται στην προσέγγιση είναι σημαντικό στοιχείο για να πετύχουμε καλύτερα τους στόχους. Όσον αφορά τις ε, αγροπεριβαλλοντικές πολιτικές που εφαρμόζονται σε ανταπόκριση στις περιβαλλοντικές πιέσεις. Νομίζω ότι κάλυψα όλες τις πτυχές ή τουλάχιστον τις σημαντικότερες που εθίγησαν. Τέλος, να υπογραμμίσω. Όταν διαβάζετε τη νέα έννοια της πολιτικής ανάπτυξης πέθρου για το μέλλον, αυτή θα εδράζεται επί έξι βασικών προτεραιοτήτων. Μεταξύ αυτών έχουμε δύο που αφορούν το περιβάλλον. Η μία με τα οικολογικά συστήματα, βάση δασοκομείας και γεωργίας, η άλλη όσον αφορά την αποδοτικότητα των πόρων. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία για να συνδεθούν με συγκεκριμένα θέματα όπως βιοπικιλότητα, Natura 2000, καλλιέργεια φιλική προς το περιβάλλον, ύδατα, διαχείριση των γεών. Αυτές οι πτυχές μαζί με καλύτερο έλεγχο, καλύτερους στόχους αποτελούν την προσπάθεια που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την πολιτική αναπτύξεως της υπαίθρου για να εξυπηρετεί καλύτερα την περιβαλλοντική διάσταση και αυτά σε συνδυασμό με τον πρώτο πυλώνα που όπως είπα θα διαθέτει 30% του προϋπολογισμού για την πράσινη διάσταση. Και στους δύο πυλώνες θα υπάρχει συμπληρωματικότητα προσπαθειών. Ελπίζω ότι το πλαίσιο ελέγχου και παρακολούθησης θα λειτουργήσει σωστά στο μέτρο για να μετράμε αποτελέσματα και συνέπειες σωστά, για να πετύχουμε τον καλό στόχο που έχουμε θέσει, που έχει θέσει η περιβαλλοντική ε, πολιτική. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και μέλη για την προσοχή σας. Ευχαριστώ Διευθυντά κύριε Σουζαούζα από την Ευθεριστική Επιτροπή για αυτά που μας είπατε. Προηγουμένως αναφέρθηκε στο Συμβούλιο. Είναι κάποιος εκπρόσωπος από το Συμβούλιο εδώ που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Φαίνεται ότι όχι. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου, τον κύριο Αλένη Σιλέ, για να ολοκληρώσει. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως είπα και προηγουμένως, υπήρχαν και βελτιώσεις στο τομέα. Το συνέδριο, το ηλεκτρικό συνέδριο δεν θέλει να υποτιμά την ε, χρησιμότητα του προγράμματος αυτού. Ταυτόχρονα θα αναφερθώ σε αυτό που είπαν οι κύριοι Ιταλα και ότι έχει φτάσει τώρα το πλήρωμα του χρόνου για να βελτιωθεί η πολιτική αυτή. Συζητείται μια νέα νομοθεσία που θα αρχίσει να ισχύει από το 2013. Και γι' αυτό ελπίζω ότι αυτή η έκθεση θα είναι χρήσιμη όταν συζητηθεί στο Κοινοβούλιο και υιοθετηθεί το νομοθετικό κείμενο για τη νέα χρονική περίοδο. Δεν θα για μια φορά να πω ότι οι συστάσεις της Κομισιόν εξασφαλίζουν διαφοροποίηση όπου κάτι τέτοιο αιτιολογείται. Και η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι πιο ενεργοί όσον αφορά την διαχείριση των πληρωμών. Να ζητούν δηλαδή από τα κράτη-μέλη να αιτιολογούν καλύτερα κατά πόσον οι στόχοι εξακολουθούν να παραμένουν ισχύοι και να χρησιμοποιούν εδώ οι βέλτες τακτικές. Η Κομισιόν έχει κάποιες προτάσεις για μετά το 2013 το λεγόμενο πρασίνισμα της κοινή αγροτικής πολιτικής. Ο κύριος Ιταλά είπε ποια είναι η συσχετισμός με αυτή την προσέγγιση. Ξέρετε, το ηλεκτρικό συνέδριο δεν είναι εκείνο που υιοθετεί την πολιτική. Αυτή τη στιγμή όμως ομολογώ ότι το ηλεκτρικό συνέδριο εξετάζει όλες τις προτάσεις της αγροτικής πολιτικής και σκοπεύουμε να γνωμοδοτήσουμε εν ευθένω 8 χρόνο βασιζόμενοι σε όλα τα αποτελέσματα που είχαμε μέχρι στιγμής. Η ευρωπαϊκή πρόταση σύμφωνα με την οποία το 30% των άμεσων πληρωμών θα σχετίζονται με κάποιες συγκεκριμένες πρακτικές αγροτικής παραγωγής είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο νομίζω της ε, πρότασης της ε, Κομισιόν. Αυτό το πρασίνισμα, αν θέλετε, ε, πλησιάζει πολύ κάποιες από τις δικές μας ε, συστάσεις. Θέλουμε δηλαδή απλούστερες και πιο απαιτητικέ δράσεις. Όπως σας είπα βέβαια δεν έχουμε καταλήξει ακόμα στην ε, προσέγγιση αυτή. Βέβαια θα μπορούσε κανένας να θέσει εδώ και το θέμα της απλούστευσης γιατί η προσέγγιση που θα υιοθετηθεί τελικά δεν θα πρέπει να αυξήσει τον πολύπλοκο χαρακτήρα και την επιβάρυνση. Εδώ θα ήθελα να κλείσω και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και την εισηγήτρια και όλη σας την Επιτροπή για την πάρα πολύ επικοδηματική συζήτηση και συνεργασία μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, για να ολοκληρώσουμε, η εισηγήτρια έχει τον λόγο. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έλαβαν το λόγο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και έδειξε πόσο σημαντική είναι η αγροπεριβαλλοντική στήριξη για τη γεωργία μας. Φαντάζομαι συμφωνείτε μαζί μου ότι τα διαθέσιμα κονδύλια για την πολιτική αυτή που ανέρχονται σε πάνω από 2 δις ευρώ θα πρέπει να δαπανώνται με το σωστό τρόπο και να συνιστούν πραγματική περιβαλλοντική αξία. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μου έδωσε ελπίδα ότι θα ληφθούν υπόψη στην πράξη τα σχόλια και οι συστάσεις μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώνουμε λοιπόν το σημείο 9 της ημερησίας διάταξης και εδώ διακόπτουμε τη συνεδρία σήμερα το πρωί. Σήμερα το απόγευμα θα συνεχίσουμε το σημείο 10 στις 3. Ευχαριστώ που προχώρησε η εργασία μας τόσο γλίγορα σήμερα το πρωί και περνάμε αμέσως και κλεισμένων των θυρών στη συνεδρία των συντονιστών.